Hello, good morning. Let's start. Καλημέρα σας, ας ξεκινήσουμε. Θα μιλήσω στα ισπανικά. Βρισκόμαστε στο σημείο 20 της ημερήσια διάταξη. Είναι η αναφορά 7 του 2018 του Αντρέ Κάουπερ, γερμανικής ηθαγένεια, σχετικά με την προγραμματισμένη αχρήστευση των λαπτήρων φωτισμού και άλλων οικιακών προϊόντων που πολλούνται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο αναφέρον δεν βρίσκεται στην αίθουσα, οπότε θα δώσω το λόγο στην Κομισιόν, στον Ρουμπέν Ντέκερ. Καλή σας ημέρα. Ευχαριστώ που μου δίνετε το λόγο. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κύριο Κάουπερ για αυτή την αναφορά που θεωρούμε ότι στηρίζει το έργο της Κομισιόν. Όπως θα είδατε από την απάντηση που έχουμε παράσχει, η Κομισιόν λειτουργεί παράλληλα, ε, εργάζεται παράλληλα σε πολλά θέματα που άπτονται αυτή τη αναφορά. Δεν θα επαναλάβω τα όσα αναφέραμε στην απάντησή μας. Αυτό μπορώ να σας δώσω σήμερα είναι μια ενημέρωση για τις τελευταίες εξελίξεις. Όπως τα διαβάσατε, ε, παίρνουμε πολύ στα σοβαρά το θέμα της επισκευασιμότητας ε, των βιομηχανικών προϊόντων στο πλαίσιο της οδηγίας Eco Design. Στην 1η Οκτωβρίου η, η Κομισιόν υιοθέτησε μια σειρά τροπολογιών ε, μέτρων της οδηγίας Eco Design για συσκευές όπως πλυντήρια, στεγνοτήρια, πλυντήρια πιάτων, ψυγεία και οθόνες μεταξύ αυτών τηλεόρασης στο όλα τα μέτρα που λάβαμε έχουμε συμπεριλάβει απαιτήσει επισκευασιμότητας. Τι σημαίνει αυτό, σημαίνει ότι όταν τα μέτρα εφαρμοστούν, οι παραγωγοί θα πρέπει να παρέχουν ανταλλακτικά για μια συγκεκριμένη περίοδο χρόνου, μεταξύ 8 και 10 ετών συγκεκριμένα, και πληροφορίες επισκευής για τους επαγγελματίες του κλάδου προκειμένου τα προϊόντα αυτά να είναι πιο εύκολο να επισκευάζονται και να επιμηκυνθεί ο χρόνος ζωής τους. Αυτό είναι ένα στοιχείο πάνω στο οποίο έχουμε συνεχίσει να εργαζόμαστε. Μια άλλη γραμμή έχει σχέση με τις προσπάθειές μας ε, να δημιουργήσουμε ένα σκορ ε, επισκευασιμότητας. Δηλαδή πόσο πολύ επισκευάσιμο είναι ένα προϊόν με έναν τρόπο ποσοτικοποιημένο. Έτσι ώστε ο παραγωγός, ο καταναλωτής, συγγνώμη, να το γνωρίζει όταν αγοράζει το προϊόν. Το Κοινό Κέντρο Έρευνας έχει εκδώσει μια τεχνική έκθεση η οποία ακριβώς εξετάζει τις πτυχές, τους παράγοντες που καθορίζουν το πόσο επισκευάσουμε ένα προϊόν. Για παράδειγμα, το πόσο εύκολο αποσυναρμολογείται, η διαθεσιμότητα ανταλλακτικών η διαθεσιμότητα πληροφοριών και για τα πιο ψηφιακά προϊόντα ε, η επικαιροποίηση του λογισμικού τους. Η έκθεση περιλαμβάνει και άλλα πράγματα, βέβαια, σας δίνω ορισμένα παραδείγματα μόνο. Αυτή τη στιγμή εξετάζουμε αυτή την έκθεση του Κοινού Κέντρου Έρευνα για να δούμε πώ θα μπορούσαμε όλε αυτέ τι πληροφορίε να τι εντάξουμε σε ένα νούμερο ε, ή ένα γράμμα, ένα σκόρ, εν πάση περιπτώσει, ε, που θα μετρά με έναν τρόπο ποσοτικοποιημένο την επισκευασιμότητα ενός προϊόντος έτσι ώστε οι καταναλωτές να το λαμβάνουν υπόψη όταν το αγοράζουν. Δύο παραδείγματα είναι αυτά από τη δουλειά που κάνουμε στην Κομισιόν. Δεν έχουμε και πολύ χρόνο, οπότε δεν θα επεκταθώ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την, τον αναφέροντα και να σα διαβεβαιώσω ότι εμεί εξακολουθούμε να εργαζόμαστε για αυτό το θέμα και θα έχουμε και συγκεκριμένα αποτέλεσματα στο μέλλον. Προεδρο, ευχαριστώ πολύ. Από τι πολιτικέ ομάδε θέλει κάποιο το λόγο. Καταρχήν, συμφωνώ πλήρω με τον αναφέροντα και, και με την ε, Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το πόσο σημαντικό είναι να είναι επισκευάσιμα τα προϊόντα στην εσωτερική αγορά για την κυκλική οικονομία και για να προστατεύουμε το περιβάλλον. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θεωρεί ότι μέχρι το 2020 ε, θα δει τους, ο κάθε λογοκυριό θα δει τους λογαριασμούς να μειώνονται κατά 500 ευρώ το χρόνο. Ε, επίσης ε, θα μειωθεί πάρα πολύ ε, η, η, το υλικό που θα χρησιμοποιείται στα προϊόντα τα οποία αγοράζουμε. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να εξασφαλίσει ότι τα προϊόντα τα οποία τη χάνουν ε, πώληση ε, θα διαρκούν περισσότερο. Επίση, πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι οι καταναλωτέ θα μπορούν εύκολα να αντικαταστήσουν, να επισκευάζουν ή να αντικαθιστούν σημαντικά ανταλλακτικά των προϊόντων του ε, και θα παράγονται περισσότερα προϊόντα τα οποία θα είναι πιο εύκολο να αποσυναρμολογούνται και να ανακυκλώνονται. Συστήνω λοιπόν να διατηρήσουμε ανοιχτή αυτή την αναφορά για να παρακολουθήσουμε τα αποτελέσματα των δημόσιων διαβουλεύσεων και να ζητήσουμε από την Κομισιόν περισσότερες πληροφορίες στο μέλλον. Σας ευχαριστώ. Δεν βλέπω να έχουμε άλλες παρεμβάσεις. Έχοντας λοιπόν εξετάσει την αναφορά και έχοντας ακούσει την Επιτροπή, θα αφήναμε ανοιχτή την εξέταση της αναφοράς αυτής, ώστε να ελέγξουμε την εφαρμογή της νομοθεσίας στα κράτη-μέλη, όπως και όλη την υπόλοιπη παρακολούθηση στην οποία προβαίνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την κυκλική οικονομία, όπως και για τον σχετικό κωδικό για την περίοδο 16-19. Να περάσουμε στο σημείο 21, που είναι η 1122 αναφορά η, από Ιταλίδα πολίτη σχετικά με τη χρήση ε, οχημάτων που έχουν εκτελονιστεί στο εξωτερικό ή εν με ε, πινακίδες κυκλοφορίας εξωτερικού, δηλαδή με ιταλικές. Οι υποβάλλοντες δεν είναι παρόντες η Επιτροπή. Έχει το λόγο ο κύριος Ρομπέρτο Μικελέτο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Εξ ονόματος της Κομισιόν να σας ευχαριστήσω για την ευκαιρία που μας δίνετε να εξηγήσουμε την κατάσταση αυτή για το ευαίσθητο αυτό θέμα, το οποίο είναι ιδιαίτερως ανησυχητικό για εμάς, για την Επιτροπή. αντιλαμβανόμαστε τα Ιταλικά μέτρα που έχουν ληφθεί και τους λόγους για τα μέτρα αυτά, διότι η διάταξη είναι υπέρ της καταπολέμησης της ε, φορολογικής απάτης και της απάτης στις ασφαλίσεις. Από την άλλη, αυτό έχει δημιουργήσει σημαντικά προβλήματα. Μάλιστα, λάβαμε αρκετέ καταγγελίε σχετικά με την εφαρμογή τη ερμοθεσία αυτή και έχουμε λάβει την πληροφορία ότι άλλε καταγγελίε υποβάλλονται μέσω άλλων υπηρεσιών. Και επομένω λαμβάνουμε το θέμα αυτό πάρα πολύ σοβαρά. Για τον λόγο αυτόν ε, έχουμε ήδη ξεκινήσει υψηλού επιπέδου επαφέ ε, και στην Επιτροπή και με τι ιταλικέ Αρχές. Το θέμα αυτό θα συζητηθεί στη Ρώμη αρχέ Νοεμβρίου σε μια σειρά συναντήσεων αφιερωμένων σε αυτό το θέμα. Είναι κάτι με το οποίο ασχολούμεθα πραγματικά και μα ανησυχεί όπως σας έλεγα πρόεδρε. Μάλιστα, ευχαριστούμε λέει ο πρόεδρος. Η κυρία Σιμαγκοπούλου. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Είναι ανισχυτική η κατάσταση στην Ιταλία, είναι σαφές. Και υπό το φως των καταγγελιών που έχουν ληφθεί, που έχουν υποβληθεί, Βεβαίω και πρέπει ούτω ή άλλω να αντιμετωπίσει το πρόβλημα τη ε, της απάτης ε, σε περίπτωση ε, ε, εκτελονισμού οχημάτων, αλλά εν πάση περιπτώσει καλό θα είναι να εξετάζουμε στενά την πορεία της αναφοράς αυτής και του προβλήματος αυτού. Ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρος. Η κυρία ε, να συμφωνήσω με τη συνάδελφο του ΕΛΚ. Είναι σαφές ότι έχουν, έχουμε λάβει καταγγελίες, αναφορές. Υπάρχει έλλειψη εναρμόνισης σε ευρωπαϊκό επίπεδο και είναι κάτι που πρέπει να παρακολουθούμε και πρέπει να μείνει ανοιχτή η αναφορά αυτή και καλό είναι να έχουμε τακτική ενημέρωση από την ε, Κομισιόν. Πολύ ωραία λέει η Πρόεδρος. Έχοντας λοιπόν εξετάσει την αναφορά, έχοντας ακούσει την Κομισιόν, έχοντας ακούσει τις πολιτικές ομάδες, η πρόταση είναι να μείνει ανοιχτή η αναφορά και να έχουμε επικαιροποιημένη ενημέρωση από την Κομισιόν προς την Επιτροπή ΠΕΤΗ, η οποία εξετάζει τις πολυάριθμες καταγγελίες που έχουν ληφθεί. Πρέπει να είμαστε ενήμεροι για κάθε νεότερο στην υπόθεση αυτή. Ευχαριστώ πολύ. Περνούμε στο σημείο 22, 1256, κάθετος 17, από τον κύριο Ραμόν Μάρκος Φερνάντεθ, Ισπανικής Μπιγκότητας, ε, εκ μέρους ε, της Ένωσης ε, Επαγγελματιών του κλάδου της αυτοκινητοβιομηχανίας σχετικά με την πρόσβαση σε πληροφορίες, σε τεχνικές πληροφορίες που είναι απαραίτητες για την επισκευή τους. Έχουμε διάφορα μέλη της Ένωσης αυτής που παρακολουθούν την εξέλιξη της αναφοράς. Θα έδινα λοιπόν το λόγο, μάλλον, στην Επιτροπή, στον κύριο Σάντσεθ Γκαλίντε, Καλημέρα σας Πρόεδρε και ευχαριστούμε πολύ τον κύριο Μάρκος Φερνάντεθ και την ε, Ισπανική Ένωση Αυτοκινητιστών για την ευκαιρία που έχουμε εδώ να παρουσιάσουμε τις τελευταίες βελτιώσεις της νομοθεσίας σχετικά με την ε, επισκευή των οχημάτων ιδιαίτερα εν ώψη του νεότερου κανονισμού του Συμβουλίου και του Κοινοβουλίου σχετικά με την πιστοποίηση, την τεχνική πιστοποίηση των οχημάτων που κυκλοφορούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ήθελα να πω ότι εμείς είμαστε απολύτως ε, ε, έτοιμοι να υποστηρίξουμε την ε, εργασία των διαφόρων οργανώσεων, διαφόρων ενώσεων που εργάζονται στο πεδίο αυτό μέσω της νομοθεσίας αυτής, του πλαισίου αυτού, η οποία αποτυπώνει τα συμπεράσματα της έκθεσης του Δεκεμβρίου του 2016 επί του πώς λειτουργεί η αγορά ως προς την πρόσβαση σε πληροφορίες σχετικές με την τεχνική συντήρηση και επισκευή των οχημάτων. Οι βελτιώσεις της νομοθεσίας αυτής, του κανονισμού, είναι οι σχετικές, τα σχετικά στοιχεία με τις ε, ε, εκπομπές, με την ασφάλεια των οχημάτων. Ε, επεκτάθηκε το σκεπτικό σε μη διακριτική πρόσβαση των κατασκευαστών εφόσον αυτοί συντηρούν τα οχήματα. Βελτιώθηκαν οι διαδικασίες επίλυσης διαφορών όταν κάποιος κατασκευαστής δεν τηρεί τις σχετικές προδιαγραφές για τη συντήρηση των οχημάτων αυτών η πρόσβαση προς τις πληροφορίες καθότι είχαμε τη διευκρίνηση ότι πρέπει αυτές να διαβιβάζονται με τρόπο αυτοματοποιημένο και ηλεκτρονικά. Υπάρχουν προϋποθέσεις λίγο πιο απλές για κατασκευαστές ειδικών οχημάτων ειδικής χρήσης Και για τα ιδιωτική χρήση οχήματα διευκρινίζεται ότι όλα τα οχήματα πρέπει να έχουν έναν, έναν OVD connector για την πρόσβαση της πληροφορίες αυτές και το, η συσκευή αυτή πρέπει να είναι διαρκώς διαθέσιμη όταν το όχημα κινείται. Ε, σε αυτή την περίπτωση μόνο για την ανάγνωση δεδομένων. Είναι από τις τελευταίες βελτιώσεις της ε, νομοθεσίας ώστε η Κομισιόν να έχει την κατάλληλη εντολή από τους συνομοθέτες ώστε να προβαίνει σε περαιτέρω βελτιώσει τη νομοθεσία και αυτό είναι που κάνουμε. Επίσης έχουμε μια σειρά προτύπων που έχουν αναπτύξει οι κατασκευαστές ε, και οι ανεξάρτητοι χρήστες σχετικά με την πρόσβαση τη πληροφορία αυτές, της συντήρησης και της ε, επισκευής. Έχουμε λοιπόν ένα νέο σχήμα πίνακα σχετικά με τις πληροφορίες για πρόσβαση σε ασφαλείς περιοχές. Η ενσωμάτωση των προτύπων αυτών αυτή τη στιγμή είναι υπό επεξεργασία και θα υποβληθεί πάρα πολύ σύντομα. Σε δεύτερη φάση η Κομισιόν θα αναπτύξει και τις υπόλοιπες τεχνικές προδιαγραφές της πρόσβασης αυτής μέσω δικτύων ε, και ώστε να υπάρχει ε, εξ αποστάσεως πρόσβαση στην τεχνική κατάσταση του οχήματο. Την εικόνα, αν θέλετε, την τεχνική του οχήματο. Ώστε να προσαρμόσουμε την νομοθεσία στις νέες τεχνολογίες που είναι διαθέσιμες πλέον για τα οχήματα αυτά. Ελπίζω υποβάλλοντες ε, να, να έχουν καλυφθεί από τις εξηγήσεις αυτές της ε, Κομισιόν, αλλά είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε πρόσθετη ερώτηση ή διαφήμιση. Μάλιστα, σε ευχαριστώ, λέει η Πρόεδρος, ο κυρία Σιμακοπούλου. Thank you, madam. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Ξεκάθαρα είναι πολύ σημαντικό για τα συνεργεία να έχουν πρόσβαση σε όλες τις τεχνικές πληροφορίες που είναι απαραίτητε για να κρατήσουν τα οχήματα σε καλή ε, κατάσταση. Το γνωρίζουμε αυτό. Και επίσης κατανοώ ότι η Επιτροπή έχει λάβει ουσιαστικά βήματα για την προσβασιμότητα σε αυτές τις πληροφορίες και τώρα επικυρωποιεί τις διατάξεις. Ευχαριστώ λοιπόν και αν δεν διαφωνεί κανείς θεωρώ ότι είναι καιρός να κλείσουμε αυτή την αναφορά. Ευχαριστώ πολύ. Είναι μεγάλη η ιστορία στην Ευρώπη για να διασφαλίσουμε τη δικαιοσύνη στον, στον ε, με τα ανταλλακτικά, να διασφαλίσουμε τους προμηθευτές ανταλλακτικών, τους κατασκευαστές, ώστε να κρατάνε τα κλειδιά ολόκληρου του τομέα. Είναι πολύ σημαντικό όσον αφορά και τους κανόνες ανταγωνισμού, τη συνεχιζόμενη προστασία και την στήριξη επίσης μικρομεσαίων επιχειρήσεων σε όλη την Ευρώπη. Ειδικά μικρά συνεργεία και γι' αυτό θεωρώ ότι είναι ένα πολύ σημαντικό αυτό το ε, θέμα αυτό που δείχτηκε από την Ισπανική Ομοσπονδία Μα είπε η Επιτροπή τι έχει κάνει ω τώρα και την ανθεώρηση των κανόνων και τα θέματα που θα αντιμετωπίσει. Επίση, τα προβλήματα που εντοπίστηκαν. Θα διαφωνήσω εδώ με τη συνάδελφα από το ΕΠΠ. Θεωρώ ότι είναι νωρί να κλείσουμε την αναφορά αυτή. Θα πρέπει να την παραπέμψουμε στην Επιτροπή Μεταφορών και στην Επιτροπή στηρικής Αγοράς, ε, καθώς είναι η υπεύθυνη επιτροπή από ό,τι βλέπω από την έκφραση του γραμματέα, αυτό μάλλον έχει γίνει. Έχει σταλεί στην ίντα. Στην Επιτροπή Μεταφορών δεν ξέρω αν έχει μεταβιβαστεί αυτή η αναφορά. Θα ήταν χρήσιμο να γίνει αυτό, γιατί είναι ένα θέμα το οποίο πρέπει να αντιμετωπιστεί, καθώς βλέπουμε ε, αυτή την ε, αλλαγή, τη μεγάλη που συμβαίνει στον ε, τομέα της κινητοβιομηχανίας ε, με τα νέα ηλεκτρονικά οχήματα που εισέρχονται στον τομέα και γενικά την εξέλιξη της τεχνολογίας. Και αυτό για να μην έχουμε αρνητικές επιδράσεις ε, στους εργαζόμενους στον κλάδο που ασχολούνται με την επισκευή. Θα πρέπει να το κρατήσουμε λοιπόν το θέμα αυτό. Ευχαριστώ την Επιτροπή για την ε, έκθεση. Θα θέλαμε να δούμε πότε θα ε, εφαρμοστούν αυτοί οι κανόνες και τότε σε εκείνη την φάση θα μπορέσουμε πλέον να κλείσουμε αυτή την αναφορά. Ευχαριστούμε κυρία Σολής. Ε, ευχαριστώ πρόεδρε. Πολύ, με πολύ ικανοποίηση παρεμένω για πρώτη φορά στην Επιτροπή ώστε να υπερασπιστώ τις οργανώσεις των αυτοκινητών. Μιλούσαμε για τους 148 εκατομμύρια καταναλωτών και στην περίπτωση Ισπανία 40.000 ε, συνολικά ε, κέντρα επισκευής με πάρα πολλούς απασχολουμένους ή η αναφορά αυτή του κυρίου Φερνάντεθ ε, μας φαίνεται θεμελιώδους σημασίας για τα κέντρα αυτά επισκευής ώστε οι καταναλωτές να μπορούν να επιλέξουν ελεύθερα την, την υπηρεσία που είναι καταλληλότερη για το όχημά τους. Πρέπει να βελτιώσουμε λοιπόν την, πρόσβαση αυτών των μικρότερη κλίμακα ε, κέντρων επισκευής στις ε, απαραίτητε πληροφορίε, ισότιμα προς τους υπόλοιπου πέκτες ε, της αγορά και ισότιμα προς τις μεγάλες επιχειρήσεις κατασκευαστών αυτοκινήτων. Θα πρέπει όμως να συγχρονίσουμε, να επικαιροποιήσουμε το συνολικό πλαίσιο, έχουμε σημαντικές τεχνολογικές πρόοδους στο πεδίο των αυτοκινήτων ε, για να είμαστε λοιπόν ανταγωνιστικοί, για να προσπίσουμε τις χιλιάδες θέσεις απασχόλησης ε, στο πεδίο, στον τομέα. Θα πρέπει η Κομισιόν να επανεξετάσει το πλαίσιο για τις σχετικές πιστοποιήσεις ανακατηγορία. Εμείς ζητούμε να παραμείνει ανοιχτή η αναφορά αυτή και οι εθνικές αρχές αποτελεσματικά και πραγματικά να ελέγχουν την ε, σχετική πιστοποίηση όλων των σχετικών κέντρων επισκευής. Ευχαριστώ πολύ. Πρόεδρος, ακούσαμε τις πολιτικές ομάδες και οπότε η πρότασή μας είναι να διατηρηθεί ανοιχτή αναφορά. Ο κυρία, κυρία Κίρτον Ντάρλινγκ έχει δίκιο έχει ήδη αποσταλεί στην ε, Επιτροπή Εσωτερική Αγοράς. Θα την ε, στείλουμε και στην Επιτροπή Μεταφορών. Διατηρούμε ανοιχτή την αναφορά. Η Κομισιόν έχει κάνει σημαντικά ουσιαστικά βήματα ε, για την διευκόλυνση της εργασίας των επισκευαστών, ε, την πρόσβαση στις πληροφορίε, ε, του τεχνικές πληροφορίες του οχήματος κλπ. Οπότε περιμένουμε όλα αυτά να υλοποιηθούν ε, έτσι ώστε ο κλάδος και οι καταναλωτές να γνωρίζουν ότι έχουμε κάνει ό,τι μπορούμε μέχρι ό,τι πραγματικά να επιληθεί το πρόβλημα ε, και να καταφέρουμε να προστατέψουμε ακόμα περισσότερο τους καταναλωτές. Ωραία. Χωρίς μικρόφωνο η πρόεδρος, δυστυχώς. Περνάμε στην αναφορά 1155 του 18 ε, ο αναφέρον είναι Πολωνός σχετικά με την απουσία ελέγχων εκπομπών οχημάτων στην Πολωνία. Ο αναφέρον απουσιάζει, οπότε θα δώσω κατευθείαν το λόγο στην Κομισιόν, στην κυρία Βίδα. Καλημέρα. Μια σύντομη ε, πληροφορία σας δώσω για την τεχνική πτυχή της αναφοράς. Ε, συνοδεύουμε από έναν συνάδελφο, ο οποίος θα συνοψίσει την πτυχή που σχετίζεται με την έγκριση τύπου οχήματο από την ε, πλευρά της Επιτροπής. Αυτό. Ο έλεγχος ε, του εξοπλισμού για τις εκπομπές ως κομμάτι του περιοδικού ελέγχου είναι κάτι που εφαρμόζεται εδώ και πολλά χρόνια. Υπάρχουν δύο καινούριε οδηγίε που εφαρμόζονται το Μάιο του 2018 και αυτές οι δύο οδηγίες έχουν εισαγάγει νέες απαιτήσει ε, για τους ελέγχους των εκπομπών για τα οχήματα Euro 5 και Euro 6 όσον αφορά την εφαρμογή αυτών των απαιτήσεων και την εποπτεία των ε, ελέγχων αυτό είναι μια αρμοδιότητα των κρατών μελών. Ο στόχος ε, για τα οχήματα ε, περιλαμβάνει και την, τον έλεγχο του ε, μηχανισμού των εκπομπών και αν λειτουργεί σωστά. Την καταλληλότητα των οχημάτων. Να κυκλοφορούν αυτό σημαίνει παράλληλα ότι όταν υπάρχει δυσλειτουργία του συστήματος ελέγχου εκπομπών, δεν παίζει ρόλο ε, στην ε, αξιοπιστία του οχήματο. Όταν δηλαδή ένα ε, εξάρτημα δεν λειτουργεί σωστά, δεν επηρεάζει απαραίτητα την καταλληλότητα του οχήματο. Κράτη-μέλη πρέπει να οργανώσουν τις δραστηριότητες τους ώστε να μπορέσουν να αντιμετωπίσουν τέτοιου είδους ε, ε, παραποιήσεις που γίνονται στον έλεγχο και αλλοιώσει και εφόσον αυτή η αναφορά αφορά την Πολωνία συγκεκριμένα, αυτό που μπορούμε να πούμε είναι ότι η Επιτροπή έχει ξεκινήσει ανταλλαγή απόψεων και ερωτημάτων όσον αφορά ε, τη διασ... Ε, αποσαφήνιση των δύο αυτών νέων οδηγιών ώστε να μην υπάρχει συστηματική παραβίαση αυτών των δύο διών Και θα δώσω τώρα τον λόγο στο συνάδελφό μου. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Από την πλευρά της έκρησης τύπου οχήματος θα πρέπει να είναι ε, συμβατά τα οχήματα αυτά που εισέρχονται στην κυκλοφορία. Είναι υποχρέωση των κρατών μελών και των κατασκευαστών να δουν κατά πόσο συμμορφώνονται ε, τα οχήματα αυτά με τις νομικές προϋποθέσεις και την οδηγία πλαίσιο και τον κανονισμό πλαίσιο. Όταν ένα όχημα παίρνει σε κυκλοφορία, είναι υποχρέωση του κράτους μέλους να εγγυηθεί ότι τα οχήματα συνεχίζουν ε, να πληρούν τις προποθέσεις ε, έγκρισης τύπου οχήματος. Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να γίνουν έλεγχοι ε, από τα κράτη-μέλη σύμφωνα με τους εθνικούς κανόνες. Δεν υπάρχουν ευρωπαϊκοί κανόνες που να ορίζουν τα τεχνικά στοιχεία που αφορούν την συνεχιζόμενη συμμόρφωση με τα πρότυπα Επίσης, σύμφωνα με τον κανονισμό, δεν πρέπει να υπάρχει αλλίωση των στοιχείων και θα πρέπει και γι' αυτό οι αρχές να κάνουν ελέγχους στη λειτουργία και θα πρέπει να γίνει και έλεγχος των εκπομπών που αυτό αποτελεί το 20% των ελέγχων. Η αλλίωση των ε, ε, συσκευών ελέγχου των εκπομπών, αυτό είναι κάτι που αφορά τα κράτη-μέλη, είναι δικιά τους ευθύνη να κρατήσουν τα όρια εκπομπών και έχει να κάνει με την ε, νομοθεσία των κρατών μελών. Ευχαριστώ κυρία Σιμακοπούλου. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Μας έδωσε το νομικό πλαίσιο η Επιτροπή σε αντίθεση με την προηγούμενη περίπτωση που είδαμε, ε, έχουμε να καλύψουμε λοιπόν μεγάλη απόσταση για να πάρουμε ξεκάθαρες απαντήσεις τόσο για την ε, εφαρμογή και εφαρμοσιμότητα αυτών των ε, οδηγιών και γι' αυτό ζητάω να μην ανοιχτή αναφορά, να διερευνήσει ακόμα περισσότερο η Επιτροπή αυτό το θέμα και για το πώς εφαρμόζεται η νομοθεσία από τις πολιτικές αρχές. Γραφεία, señora Κίρτον. Um, yes. Ε, ναι. Ε, συμφωνώ με τη συνάδελφό μου από το ΕΛΚ. Θεωρώ ότι ένα επιπλέον σημείο είναι ότι εμείς θέτουμε ένα πλαίσιο για μια ζωτική σημασίας νομοθεσία. Αν αναλογιστούμε και το, την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής είναι ένα πολύ ε, μεγάλη σημασία θέμα αυτό για την Ευρωπαϊκή Ένωση και γι' αυτό η ιδέα ότι νομοθετούμε για ισχυρότερους ελέγχους αλλά όταν ε, κάποιος οδηγεί υπάρχουν αλλοιώσεις στις εκπομπές οπότε παραβιάζεται αυτή η νομοθεσία τότε θα πρέπει να ανισχύσουμε για αυτό το θέμα. Συμφωνώ με την αδελφό από την ΕΛΚ. Ακούσαμε ποιο είναι το νομοθετικό πλαίσιο. Όπως και οι περισσότερες αναφορές μας, ε, αυτή η αναφορά έχει να κάνει με την εφαρμογή, πώς εφαρμόζονται οι οδηγίες στα κράτη-μέλη. Γι' αυτό θα θέλαμε περισσότερες πληροφορίες για να δούμε τι συμβαίνει στην Πολωνία σε σχέση με τις εκπομπές. Γι' αυτό θέλουμε να μην ανοιχτή αναφορά και θα θέλουμε να εμβαθύνει στο θέμα περισσότερο η Επιτροπή και να επανέλθουμε περισσότερες πληροφορίες και οι δύο ομάδες που μίλησαν ζήτησαν να μείνει ανοιχτή η αναφορά. Αυτό προτείνω και εγώ, όπως και η κυρία Κίρτον, όπως και η κυρία Σιμακοπούλ, να πω ότι η Κομισιόν κατέστησε σαφές ότι η νομοθεσία απαγορεύει ρητά ε, την ε, τροποποίηση των τεχνικών χαρακτηριστικών των οχημάτων, την παραποίησή τους, ε, και τα κράτη-μέλη θα πρέπει να την εφαρμόζουν αυτή την νομοθεσία. Ε, οπότε σε αυτά ε, πέφτει το βάρος από το 2020 και μετά. Τα κράτη-μέλη θα πρέπει να κάνουν τακτικούς ελέγχους έτσι ώστε τα κυλοφορούν τα οχήματα, τηρούν τις νομικές προδιαγραφές και τις νομικές απαιτήσει. Οπότε αυτό που θα πρέπει να συνεχίσουμε να κάνουμε εμείς είναι να, να, να βεβαιωνόμαστε ότι θα εξακολουθεί να εφαρμόζεται η Ευρωπαϊκή Νομοθεσία αφενό και φετέρου, από το 2020 και μετά να είμαστε σίγουροι ότι τα κράτη-μέλη πραγματικά θα ξεκινήσουν αυτού του τεχνικού ελέγχου. Ε, Πάντω η νομοθεσία ήδη έχει υιοθετηθεί, έχει μεταγραφεί και θα πρέπει να αρχίσει να εφαρμόζεται από το επόμενο έτο. Ευχαριστώ πολύ. Περνάμε στο σημείο 24. Αναφορά 1116 του 18 του Αντώνιο Εσκόβαρ, Εσκοβάρ Φλόρεθ, Ισπανική Σταγένεια, εξ ονόματο τη ε, το Ανεξάρτητο Σωματείο Πληρώματο Θαλάμου Επιβατών, σχετικά με τι παραβάσει τη νομοθεσία από τη Ryanair στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι εδώ ο αναφέρον. Καλώ ήρθατε. Έχετε πέντε λεπτά, κύριε Σκομπάρ, για να μας παρουσιάσετε την αφορά σας. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Καλή σας μέρα. Θα προσπαθήσω να είμαι όσο πιο σύντομος γίνεται. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει ένα συνολικό σχέδιο έτσι ώστε η Ryanair να εφαρμόζει την νομοθεσία ε, και να αναλάβει τις κοινωνικές ευθύνες. Η Ryanair εκμεταλλεύεται τα παράθυρα της νομοθεσίας να τα οποία οδηγούν, την επιτρέπουν μάλλον να καταχράτε τα δικαιώματα. Ε, η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να πάρει τα αντίστοιχα νομοθετικά μέτρα. Ε, δεν θα πρέπει να έχουμε σημαίες ευκαιρίες στην, ευκαιρίας στην Ευρωπαϊκή αεροπλοία. Η Ryanair έγινε μια μαγική, ένα μαγικός αερομεταφορέας με ρυθμούς ανάπτυξης τεράστιους. Σύμφωνα ε, με μελέτες που έχουν γίνει, αν η Ryanair ε, πλήρωνε όλες τις κοινωνικές φορές που θα έπρεπε και λοιπά, θα κέρδιζε 20% λιγότερο. Δηλαδή η λειτουργία της Ryanair είναι μια απάτη. Αυτή η απάτη όμως για τα πληρώματα είναι ένας εφιάλτης καθημερινά. 20.000 οικογένειες ε, ζουν σε αυτή την ε, νεκρή ζώνη του νόμου, όπως την αποκαλούμε, ε, και υφίστανται πολύ κακή συμπεριφορά. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση όμως όλοι είμαστε ίσοι. Θα ήθελα να σας ζητήσω να απαιτήσετε από τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης να, τους, ε, να σας δείξουν τις εκατοντάδες δικαστικές αποφάσεις εις βάρος της ΡΑΕΝΕΡ που την καθιστούν ε, πειρατή των εθέρων. Ε, οι επιθεωρητές εργασίας, ε, δικαστές, ε, εθνικές διοικήσεις κλπ. μας δίνουν δίκιο. Τι κάνουν όμως οι εθνικές κυβερνήσεις. Με την εξαίρεση της Γερμανίας, οι υπόλοιπε ε, χώρες αποφάσισαν ε, να ε, κλείσουν τα μάτια. Έχει έρθει όμως η ώρα, η μεγάλη πλειοψηφία των αεροπορικών εταιριών, των αερομεταφορέων, να τύχουν του σεβασμού που χρειάζονται. Θα πρέπει, γιατί βρίσκονται σε μειονεκτική θέση. Γιατί, Γιατί αυτές σέβονται την εθνική Νομοθεσία και την ευρωπαϊκή νομοθεσία. Η ε, απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου, η υπόθεση Μόνς του 2017, ε, ε, ήρθε 8 χρόνια μετά την πρώτη καταγγελία των πληρωμάτων του Ryanair, της Ryanair και τελικά δεν χρησιμεύσε και σε τίποτα. Ε, θα πρέπει όμως η Ευρωπαϊκή Ένωση να λειτουργεί ε, υπέρ των πολιτών. Και η Ρώμα 1 και η Βρυξέλλες 1, οι δύο συμβάσεις δηλαδή, θα πρέπει να λειτουργούν και να εφαρμόζονται πλήρως. Εφόσον έχουν ληφθεί αρνητικές αποφάσεις για τη ΡΑΕΝΕΡ, θα πρέπει να λαμβάνονται και προστατευτικά προληπτικά μέτρα. Γιατί η δικαιοσύνη αργεί. Και οι εθνικέ και οι τοπικέ κυβερνήσει στην Ισπανία, για παράδειγμα την Πολώνια και την Πορτογαλία, χρηματοδοτούν ή βοηθούν οικονομικά ε, αυτούς ε, τη Ryanair. Θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση να πάρει μέτρα. Δεν είναι δυνατόν να δίδονται παραπάνω σλότ στην Ryanair μέχρι σότου ε, πληρεί τα ελάχιστα τουλάχιστον, τις ελάχιστα τουλάχιστον κοινωνικές και ε, επιχειρηματικές προδιαγραφές. Γιατί, γιατί άλλες αεροπορικές εταιρείες θα τη μιμηθούν. Ε, η προσβολή στα εργατικά, εργασιακά δικαιώματα έχουμε, ε, γίνεται με πολλούς τρόπους. Στην ε, Πολωνία γίνεται κάτι τρομακτικό. Το 2009 απέστειλε μια, ένα επιστολή στα πληρώματα με, εκβιάζοντας τα πληρώματα να λειτουργούν ως ψευδοαπασχολούμενοι γιατί αλλιώς θα απολυθούν. σε αυτή την περίπτωση ποιος θα ε, αποζημίωνε τα θύματα. Ε, στην Τσεχική Δημοκρατία και στη Βουλγαρία τα πληρώματα έπήραν μια επιστολή που τους λέει ότι από τις 27 ή θα ε, υπογράψεις με την Ryanair Bus ή αλλιώς θα απολυθείς. Στην Ισπανία δεκάδες καταγγελίες οδήγησαν σε επιθεωρήσεις Ρασίας που οδήγησε σε πρόστιμα τη Ryanair για προσβολή των δικαιωμάτων απεργίας ε, και διαρκή κατάχρηση ε, εξουσίας. Στην Ισπανία και την Πορτογαλία ε, γίνεται παρερμηνία των εθνικών, της εθνικής νομοθεσίας περί ελάχιστων, ελάχιστων πληρωμάτων σε μέρες απεργίας. Όμως οι κυβερνήσεις αυτές είναι συνένοχες διότι ε, επιτρέπουν απεργίες ε, με μηδενικές ακυρώσεις πτήσεων. Με αυτόν τον ε, τρόπο επιβάλλουν, η Ryanair επιβάλλει ψευδοσυμβόλαια μηδενικών ορών εργασίας, μεταφέρει πληρώματα από τη μία χώρα σε άλλη για να αντιμετωπίσει απεργίες κλπ. κλπ. Στην holding Ryanair υπάρχουν ε, ψευδο αερομεταφορείς βιτρίνες ε, με τρόπο ώστε να παρακάμπτονται τα δικαιώματα των πληρωμάτων. Δεν είναι όμως μόνο εργασιακό το θέμα. Από τη Βαρκελόνη, ας πούμε. Η Ryanair κάθε εβδομάδα, για παράδειγμα, εισπράττει 50.000 ευρώ. Αυτά τα 50.000 πάνε σε σάκους στο Δουβλίνο. Πώς ελέγχονται, ποιο ελέγχει αυτές τις μεταφορές ποσών. Ε, δεν θα έπρεπε πάνω από 10.000 να ελέγχονται. Παρακαλώ πολύ λίγο πιο αργά, διότι οι διερμηνείς θα πρέπει να μπορούν να μεταφράζουν και αυτοί κανονικά, γιατί μιλάτε πάρα πολύ γρήγορα. Το σημαντικό είναι να μεταφράσετε και σωστά για να σας καταλάβουν. Λέω λοιπόν, εισπράττονται 50.000 ευρώ μία εβδομάδα ε, για τις πτήσεις από τη Βαρκελόνη. Ε, αυτά τα 50.000 ευρώ ε, πηγαίνουν στο Δουβλίνο σε σάκους στο Δουβλίνο. Πού φορολογούνται, Ποιο ελέγχει αυτέ τι μεταφορέ, τι γίνεται με την εθνική νομοθεσία που υποχρεώνει να ελέγχονται μεταφορέ ποσών πάνω από 10.000 ευρώ. Η Ryanair αποφεύγει τις κοινωνικές ε, εισφορές και ταυτόχρονα στέλνει χρήματα με αεροπλάνο και σάκους από τη μία χώρα σε μία άλλη ε, είναι μια επιχείρηση πολύ προβληματική για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι τεράστια. Δεν, μπορεί να, ε, δεν μπορούμε προφανώς να την κλείσουμε. Αλλά πρέπει να σέβεται την νομοθεσία. Γιατί αυτή τη στιγμή ε, αντιπροσωπεύει μια ελίτ, επιχειρηματική ελίτ, μια επιχειρηματική αριστοκρατία που ζει στο περιθώριο του νόμου και κανένας δεν μπορεί να την ακουμπήσει. Στην Ιταλία, τη Γαλλία και τη Γερμανία η Ryanair ανακοίνωσε μια, ένα rebranding γιατί έχει καεί ως όνομα ή μια καινούρια ε, ε, η Malta Air που είναι μια καινούρια ένας καινούριος αερομεταφορέας του, της ομάδας αυτής του ομίλου ε, αναλαμβάνει όλη τη λειτουργία της Ryanair σε αυτές τις χώρες είναι όμως μια ένας αερομεταφορέας από μια πολύ μικρή χώρα, κάτι που θα οδηγήσει σε ακόμα μικρότερη, μικρό, λιγότερο έλεγχο και λιγότερες επιθεωρήσεις. Τελειώνω λέγοντας ότι η ελευθερία της ενιαίας αγοράς είναι καλή, απαραίτητη και ο ανταγωνισμός μας βελτιώνει. Όμως είναι απαράδεκτο ε, χάρη σε αυτή την ελεύθερη αγορά να γίνονται τέτοιες προσβολές στα εργασιακά δικαιώματα και θα πρέπει να πάρουμε την κατάσταση στα χέρια μας. Σας ζητώ λοιπόν το Κοινοβούλιο να απαιτήσει από τα κράτη-μέλη μια έκθεση που να περιγράφουν τις πραγματικές δράσεις, πράξεις κυβέρνηση έτσι ώστε η Ryanair να τηρεί την νομοθεσία και βέβαια τις συμφωνίες που έχουν υπογράψει με τη Ryanair σε κάθε χώρα. Θα έπρεπε να έχουμε ένα benchmark, ένα κανόνα με βάση τον οποίο να μπορούμε να συγκρίνουμε τις λειτουργίες και τη δράση των αερομεταφορέων έτσι ώστε να μην έχουμε στο μέλλον απεργίες με μηδενικές ακυρώσεις. Η... Ας... Ας ζητηθεί από την ε, ETF έτσι ο, ε, να ζητηθεί από την ETF να συνεργαστεί έτσι ώστε αυτό το καθεστώς προβλέπεται για τους ε, ε τα αυτοαποσχολούμενα πληρώματα της οδηγίας 2008-2008 ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης να γίνει πραγματικότητα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστούμε εμείς λέει η Πρόεδρος. Η κυρία Ντελαβαρέρο Φλόρεθ από πλευρά τη Κομισιόν έχει λόγο. Σα ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ακούγοντα τον υποβάλλοντα, δεν μπορώ παρά να θυμίσω την ε, παρέμβαση του Πρόεδρου Γιούνκερ εδώ, σε αυτόν τον οίκο, το 2016, όταν αναφερόμασταν στο γεγονό ότι ούτε η Ευρωπαϊκή Ένωση, ούτε ο αεροπορικός της χώρος δεν είναι η Άγρια Δύση. Έχουμε δίκαιο, εφαρμόζεται από τα κράτη-μέλη. Πρέπει λοιπόν όλοι οι οικονομικοί φορείς να τηρούν τις διατάξεις, την νομοθεσία, την ευρωπαϊκή και την εθνική. Εγώ συμφωνώ με την βασική γραμμή της αναφοράς που αναφέρεται στην σωστή εφαρμογή της νομοθεσίας στα διάφορα κράτη-μέλη αυτή τη φορά από πλευράς συγκεκριμένης επιχείρησης. Αυτό αφορά και στα εργασιακά και κοινωνικά δικαιώματα. Αναφέρθηκε στον ε, κανονισμό Ρώμη 1 και Βρυξέλλες 1 ο υποβάλλοντας και αυτό αναφέρεται και εδώ στην σωστή εφαρμογή της νομοθεσίας από πλευράς τη επιχείρησης. Εξαρτάται λοιπόν από τις αρχές των κρατών μελών και ιδιαίτερα της Ισπανίας σε αυτή την περίπτωση να τηρούν, να εφαρμόζουν την νομοθεσία αυτή και να υποχρεώνουν τις επιχειρήσεις να την τηρούν. Η Κομισιόν έχει αναλάβει απόλυτη δέσμευση να προστατεύει όλους τους εργαζομένους, ιδιαίτερα στο πεδίο των αερομεταφορών. Και γι' αυτό ενεκρίθηκε μια έκθεση στις αρχές του έτους, το Μάρτιο, για τις κοινωνικές επιτυχίες της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής ε, για τις αερομεταφορές και εκεί είχαμε υποδείξει διάφορες κατευθύνσεις, ε, επίπεδα στα οποία μπορούσαμε να υποστηρίξουμε τα κράτη-μέλη, καταρχάς τους κοινωνικούς φορείς μέσω του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Διαλόγου, στην Επιτροπή της ε, Πολιτικής ε, Αεροπορίας συγκεκριμένες επιχειρήσεις, όπως η Ryanair, ε, σημειώθηκαν στο τελευταίο συνέδριο μεταξύ των κοινωνικών φορέων. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε κάθε περίπτωση είναι δεσμευμένη να υποστηρίζει τα κράτη-μέλη ώστε να εφαρμόζονται οι διατάξεις. Ε, μιλούμε για ένα τομέα όπου έχουμε υψηλότατη κινητικότητα, έχουμε διάφορες, αν θέλετε, τεχνικές δυσκολίες σχετικά με αυτό, αλλά γι' αυτό προσπαθούμε να συστήσουμε μια ομάδα εμπειρογνωμόνων των κρατών μελών αεροναυπηγικής και εμπειρογνωμόνων των Υπουργείων Εργασίας ε, και Κοινωνικής Ασφάλισης, ώστε να παρακολουθούμε τις εξελίξεις στο θέμα αυτό και τις βασικότερες πτυχές στις οποίες αναφέρθηκε και ο υποβάλλοντας, δηλαδή αυτούς που εμφανίζονται ως ελεύθεροι επαγγελματίες ενώ δεν είναι, ε, και άλλες περιπτώσεις παραβίασης ή παράκαμψης των διατάξεων του εργασιακού δικαίου. πρέπει να τηρούμε υψηλά πρότυπα προστασία ε, των εργαζομένων σε όλες τις χώρε τη Ευρωπαϊκή Ένωση και πρέπει να συνεχίσουμε να ενισχύουμε τα κράτη-μέλη, ιδιαίτερα στις αεραμεταφορές. Ευχαριστούμε. Yes, thank you, Chair. Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Και ο και εγώ από την ε, που συμμετέχω στην Επιτροπή Επασχόληση. Είναι πολύ σημαντικό το θέμα αυτό που έθιξε ο αναφέρον, καθώς βλέπουμε πολλά ε, παραθυράκια στο νόμο που επιτρέπουν την παραβίαση. Το, την έννοια της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως μια κοινωνική ένωση για να εκπληρώνει τις υποχρεώσεις της έναντι των εργαζομένων. Αυτό που θα ήθελα να πω ε, στον εκπρόσωπο της Επιτροπής κάνετε λόγο για να εξετάσουμε την παραβίαση της τρέχουσας νομοθεσίας, αλλά είναι προφανώς ότι θα πρέπει αυτά τα νομικά παραθυράκια να εξαλειφθούν μέσα, μέσω βελτίωσης της νομοθεσίας Ακούσαμε τον αρμόδιο επίτροπο, ο οποίος υποσχέθηκε να αναλάβει πρωτοβουλία όταν ανακαλυφθούν ε, αυτά τα νομικά παραθυράκια. Τα παραθυράκια αυτά εντοπίστηκαν πλέον η ΡΑΙΝΕΡ δημιουργεί πρόβλημα με τις ε, συμβάσεις ε, που παρέχει στους εργαζόμενους και δεν τους εξασφαλίζει, δεν ε, τους παρέχει την απαραίτητη, την προβλεπόμενη ασφάλιση. Θα πρέπει λοιπόν να υπάρξουν τροπολογίες στην νομοθεσία. Και η πρότασή μου είναι η εξή. Επίση, να πω ότι είναι πολύ καλό που ε, την ομάδα εμπειρογνωμόνων, η οποία θα μπορέσει να προτείνει ε, νομοθεσία. Θα ήθελα λοιπόν να προτείνω να κρατήσουμε την αναφορά αυτή ανοιχτή. Να στείλουμε τις πληροφορίες της Επιτροπές Απασχόλησης ε, και Μεταφορών και να ζητήσουμε από την Επιτροπή να είναι πιο δραστήρια στις προτάσεις ε, αυτές για νέα νομοθεσία. Σαλίβα. First of all, I would like to thank the... Ο κύριος Σαλίβα, να ευχαριστήσω τον υποβάλλοντα που ε, ε, έθεσε αυτό το πολύ σημαντικό θέμα των παραβιάσεων από πλευρά της Ryanair. Δεν είναι η πρώτη φορά που ασχολούμαστε με τέτοιου είδους περιπτώσεις και πρέπει να εξακολουθούμε να ασκούμε πίεση στην Ryanair για τα πληρώματα θαλάμου που είχαν φτάσει σε ένα σημαντικό σημείο ώστε να προστατεύσουν τα κοινωνικά συστήματα ασφάλισης για τα μέλη του πληρώματος θαλάμου που είναι ε, πολύ σημαντικό για το πρότυπο της ε, εργασίας και της κοινωνικής ασφάλειας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Εγώ θα ζητούσα από την Πρόεδρο να, να κρατήσουμε την αναφορά ανοιχτή και να παρακολουθεί η Κομισιόν την ε, μετεγγραφή των διατάξεων ε, εργασιακού δικαίου και κοινωνικού δικαίου προς την Ισπανία ιδιαίτερα ως προς τη Ryanair. Ευχαριστούμε κυρία Μαέστρε. Ευχαριστώ πρόεδρε. Πρώτα απ' όλα να ευχαριστήσω τον κύριο Εσκοβάρ που ήρθε εδώ να μας παρουσιάσει αυτό το θέμα που είναι πάρα πάρα πολύ σημαντικό και δεν είναι η πρώτη φορά που μας απασχολεί. Γιατί δυστυχώς η Ryanair καθίσταται περιβόητη σιγά σιγά. Με διάφορες τέτοιες περιπτώσεις καταγγελιών είχαμε για πριν από ένα μήνα ή κάτι τέτοιο που, από Ένωση Καταναλωτών της χώρας μας που κατήγγελε τις ε, παραβιάσεις ε, που, στις οποίες ε, διαρκώς τακτικά προβαίνει η επιχείρηση αυτή. Παραβιάσεις του εργασιακού και του κοινωνικού δικαίου είναι σίγουρο ότι η έκθεση στην οποία αναφέρθηκε η Κομισιόν και διάφορα μέσα που έχει διάθεσή τη μπορεί να τα χρησιμοποιήσει πιο αποτελεσματικά. Εδώ έχουμε να κάνουμε μια επιχείρηση που δρά διεθνώς, οπωσδήποτε διασυνοριακά και οπωσδήποτε αφορά άμεσα και στη χώρα μας. Και πρέπει οι εθνικές αρχές να συμμετάσχουν ε, και σε διεθνές επίπεδο και σε εθνικό επίπεδο. Έχουμε στη διάθεσή μας λοιπόν μέσα τη επιτροπή. έχουμε μέσα εμείς εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ως Επιτροπή Πέτη, ε, με, με την Επιτροπή Μεταφορών, με την Επιτροπή Απασχόλησης, πρέπει όχι μόνο να διατηρήσουμε ανοιχτή την αναφορά αυτή, αλλά να κοιτάξουμε να σχηματίσουμε, να συστήσουμε μια ομάδα εργασίας ώστε να έχουμε διαρκή ενημέρωση σχετικά με τις σχετικές εκθέσεις και να έχουμε μια κοινή δράση αντιμετώπισης του πολύ αυτού. Αν δεν κάνω λάθος, ε, μάλιστα ε, ανακοινώθηκε ο πλευράς ε, της επιχείρησης αυτής ένα δισεκατομμύριο τιμολόγηση έχει το περασμένο έτος η επιχείρηση αυτή μόνο στην Ισπανία, μόνο στην Ισπανία, και τις εισπράξεις αυτές είναι η τρίτη πηγή εσόδων είναι η χώρα μας, αντιπροσωπεύει για την επιχείρηση αυτή ε, και αφορά και πάρα πάρα πολλούς εργαζομένους. Δεν μπορούμε να περιμένουμε, δεν μπορούμε να καθυστερούμε. Πρέπει αυτή η επιχείρηση ε, ούτε να εκμεταλλεύεται, ούτε να εκβιάζει τη χώρα μας ή οποιαδήποτε άλλη χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ούτε να παραβιάζει τις διατάξεις νομοθεσίας. Και όπως είπαν και οι συνάδελφοι της Επιτροπής, θα πρέπει να επικαιροποιήσουμε τέλος πάντων την απάντησή μας, την ανταπόκρισή μας. Σας ευχαριστώ. Ο κύριος. Ευχαριστώ. Σε πολλές άλλες περιπτώσεις θα υποστήριζα την ε, ευελιξία στην εργασία. Όταν όμως αφορά ύψιστα θέματα ασφαλείας, όπως είναι με τα πληρώματα καμπίνας, η ευελιξία δεν έχει χώρο. Η ασφάλεια, η συνεργασία είναι πιο σημαντική. Επομένως θεωρώ ότι και η αναφορά και τα αποτελέσματα που μας έδωσε η Επιτροπή είναι πολύ σημαντικά. Θα πρέπει να μην ανοιχτή η αναφορά, τουλάχιστον μέχρι να υπάρξει μια πιο σταθερή νομοθετική απόφαση. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε δεν είναι δυνατόν να μην ε, αντιδρούν οι αρχές και να δείχνουμε και ανοχή σε κατάσταση, σε μια καταπάτηση εργασιακών δικαιωμάτων που θέτει επίσης σε κίνδυνο και την ε, ασφάλεια των αερομεταφορών. Γι' αυτό και η δικιά μας η ομάδα ζητά να μείνει ανοιχτή η Επιτροπή για περισσότερες πληροφορίες και να φτάσουμε σε, μια, σε ένα αποτέλεσμα. Ευχαριστώ. Thank you. Uh, señor Nicolai Alavanos. Ο κύριος Αλαβάνος. Gracias, Presidenta. Ε, εγώ hablar en griego. Ε, άκουσα μεγάλη προσοχή την αναφορά που έφερε στην προσοχή της Επιτροπής μας ο Ετών, ε, όπως και τα σχόλια της εκπροσώπου της Κομισιόν και την αιτιολόγηση που έχει κάνει η Κομισιόν. Ε, Αρχικά πρέπει να πούμε ότι είναι μια πάρα πολύ ολοκληρωμένη και μελετημένη ε, αναφορά που παρουσιάζεται και σε σχέση με τα μέτρα που πρέπει να παρθούν. Πράγμα το οποίο είναι πάρα πολύ σοβαρό με την έννοια ότι δίνει και μια κατεύθυνση. Θέλω να υπογραμμίσω το εξή ζήτημα. Βεβαίω η συγκεκριμένη εταιρεία πάρα πολλέ φορέ έχει απασχολήσει. Ε, Όμω, όπω είπαν και προηγούμενοι, το πλαίσιο το οποίο ε, υπάρχει ήδη, το οποίο επιτρέπει την υπερεκμετάλλευση και τη διάλυση των εργασιακών σχέσεων και των πληρωμάτων των αεροπορικών εταιριών, των πληρωμάτων καμπίνας, εκεί οδηγεί. Είναι <clears throat> υποκριτικό, κατά την άποψή μας, από την πλευρά της Κομισιόν, τη στιγμή που σε δεκάδες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης προωθούνται μέτρα τα οποία χτυπούν το δικαίωμα στο συνδικαλισμό, το δικαίωμα στην απεργία, χτυπούν το δικαίωμα στις συλλογικέ συμβάσεις εργασίας, στην ύπαρξη σταθερής και μόνιμης εργασίας, να θεωρούμε ότι σε αυτό το πλαίσιο θα έρθει η Κομισιόν και θα επιβάλλει με αυτόν τον τρόπο στις ιδιωτικές επιχειρήσεις ε, του κλάδου της, των αερομεταφορών αυτή την κατάσταση. Εμείς συμφωνούμε να μείνει ανοιχτή η αναφορά. Χρειάζεται με κάθε μέσο που έχουμε στα χέρια μα να πιέσουμε έτσι ώστε να λυθούν αυτέ οι ακραίε καταστάσεις που δημιουργούνται, όμως γνωρίζουμε ότι δεν υπάρχει άλλη λύση πέρα από τον οργανωμένο συλλογικό αγώνα των εργαζομένων, έτσι ώστε να μπορέσουν να κατακτήσουν τα δικαιώματά τους. Και σε αυτή την κατεύθυνση θα μας έχουν ε, στο πλάι τους. Ευχαριστώ πολύ. Muchísimas gracias. Ahora, como no hay más intervenciones para finalizar este punto. Σας ευχαριστώ. Ε, ώστε να ολοκληρώσουμε το σημείο αυτό και πάλι ο κύριος Εσκοβάρ έχει δύο λεπτά για να κλείσουμε το σημείο σας παρακαλώ. Ευχαριστώ Πρόεδρε, ευχαριστώ όλους τους ε, παρεμβαίνοντες. Θα επαναλάβω τα λεγόμενα της ε, εκπροσώπου της ε, Κομισιόν. Δεν είναι η Άγρια Δύση, δεν είναι το Φαρουέστ αυτό. Είναι σημαντικό να έχουμε μια συλλογική συνειδητοποίηση ότι η ευρωπαϊκή νομοθεσία, η ενωσιακή νομοθεσία είναι πλήρης, είναι καλή, καλύπτει τι περισσότερε περιπτώσει και είναι καλή για του περισσότερου εκτό από τη Ryanair. Πρέπει να παρακολουθούμε τη δράση τη εταιρεία αυτή. Στη Γερμανία ε, νομίζω ότι έχουν καταφέρει να επιβάλλουν τις διατάξεις νομοθεσία. Ε, στη χώρα μα όχι, πρέπει να γίνει. Σα ευχαριστούμε κύριε Σκοβάρη, λέει η πρόεδρο, που ήρθατε εσείς προσωπικά να μας παρουσιάσετε την αναφορά σας έχοντας ακούσει εσάς την Κομισιόν, τις πολιτικές ομάδες, θα πρότεινα καταρχάς να διατηρήσουμε ανοιχτή την αναφορά και να αποστείλουμε μία επιστολή στη Ryanair, μία ενημέρωση, ώστε να γνωρίζει τις διάφορες αναφορές που έχουν υποβληθεί, τις καταγγελίες των καταναλωτών και των απασχολουμένων της, των εργαζομένων της, και θα αποστείλουμε επίσης επιστολή στις Ισπανικές αρχές, αλλά όχι μόνο σε αυτές που αναφερθήκατε εσείς, τις εργασιακές, ε, τις αρχές κοινωνικής ασφάλισης, τις ε, πολιτικής αεροπορίας, για τις συγκεκριμένες ε, παραβιάσεις στις οποίες αναφερθήκατε, ώστε να υποστηρίξουν και το διάλογο μεταξύ των εκπροσώπων των κοινωνικών, των των διαφόρων εργαζομένων τη εταιρεία και όχι μόνο στην Ισπανία αλλά σε όλες τις χώρες που δραστηριοποιείται η εταιρεία αυτή ώστε να είναι όλοι ενημερωμένοι σχετικά με τις διατάξεις της ε, νομοθεσία σε όλες τις χώρες αυτές και που πρέπει να εφαρμόζονται από την επιχείρηση, από την εταιρεία. Μέσω τη επιτροπή Μεταφορών, αναφορών με συγχωρείτε, θα, θα ενημερώσουμε και την Επιτροπή Κοινωνικών Θεμάτων και την Επιτροπή Μεταφορών για τα όσα ακούσαμε εδώ και θα ζητούσαμε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ευχαριστώντας ε, τους συναδέλφους για τη δουλειά που κάνουν στο επίπεδο αυτό θα πρέπει να εξακολουθήσουμε να ε, αναζητούμε λύσεις για τα προβλήματα των εργαζομένων που εμφανίζονται ως ελεύθεροι επαγγελματίες μεταξύ άλλων, ώστε και το, συνολικά το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να μπορεί να, έχει, να διατηρεί ε, την πρωτοβουλία του και την προσπάθειά του να προστατεύει τους καταναλωτές και τους εργαζομένους όλων των επιχειρήσεων και στην συγκεκριμένη περίπτωση βεβαίω της Ryanair. Σας ευχαριστούμε για την αναφορά σας. Να προχωρήσουμε στο σημείο 25. 393 κάθετος 2013 από Βρετανό υπήκο με 750 υπογραφές για τη νέα ισπανική νομοθεσία σχετικά με την υποχρέωση ε, Υποβολή των στοιχείων ενεργητικού, των περιουσιακών στοιχείων και δικαιωμάτων που κατέχει κανεί στο εξωτερικό μαζί με την 478 και 566 από τους ε, Πα, Πατρίκ Λεκάμ και Άντο Ριβάλκε σχετικά και πάλι με την Ισπανική νομοθεσία για την υποχρέωση ε, αναφοράς των ε, περιουσιακών στοιχείων και δικαιωμάτων που κατέχονται στο εξωτερικό και της 073815 και πάλι για την κατοχή περιουσιακών ε, στοιχείων ή συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων στο εξωτερικό. Θα έδινα το λόγο σε δύο από τους εκπροσώπους, σε έναν, μου λένε. Α, στον κύριο Βάλκε. Παρακαλώ, πέντε λεπτά, έχετε το λόγο. Thank you very much, Madam Chair. Uh, good morning. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Είναι χαρά μου που βρίσκομαι και σήμερα εδώ. Ευχαριστώ που μας ξανακαλέσετε για να συζητήσουμε αυτή την αναφορά Υποβλήθηκε πρώτη φορά το 2013 και αφορά την υποχρέωση υπό ισπανικό δίκαιο να υποβάλλονται στοιχεία για κατοχή περιουσίας εκτός Ισπανίας. Δεν αφισβητούμε την υποχρέωση να δηλώνουν ε, τα περιουσιακά του στοιχεία. Αυτό που μας προβληματίζει είναι η αναλογικότητα των μέτρων, γιατί υπάρχουν διακρίσεις που γίνονται όσον αφορά την υποχρέωση την υποχρέωση υποβολής ε, φορολογικής δήλωσης. Υπάρχει διακριτική μεταχείριση για ε, περιουσιακά στοιχεία που έχει κάποιος στην Ισπανία και άλλο που έχει στο εξωτερικό. Για τα περισσότερα στοιχεία στο εξωτερικό είναι πιο, θα λέγαμε, δεσμευτικές και αυστηρές υποχρεώσεις. Σύμφωνα ε, με τις φορολογικές υποχρεώσεις ε, για περισσότερα στοιχεία εκτός εξωτερικού, οι προθεσμίες υποβολής είναι πιο σύντομες, οι κυρώσεις ε, για καθυστέρηση είναι υψηλότερες. μέχρι και 10.000 ε, ευρώ μπορεί να είναι τουλάχιστον το πρόστιμο για ελλειπή υποβολή στοιχείων. Και 200 ευρώ για υποβολή περιστικών στοιχείων που ε, αφορούν ε, περιουσιακά στοιχεία στην Ισπανία. Υπάρχει λοιπόν μια δυσαναλογία και περιλαμβάνονται και οι επενδύσεις σε άλλες χώρες όπου και πάλι οι υποχρεώσει είναι υποβολής ε, στοιχείων είναι πιο ε, δεσμευτικέ. Είμαστε πολύ ικανοποιημένοι με την Επιτροπή που μετά από έρευνα αποφάσισε να παραπέμψει το θέμα στο δικαστήριο. Και επίσης ήθελα να τονίσω ότι προφανώς τα μέλη θα είναι στη θέση να διακρίνουν ότι το επίπεδο ενασχόλησης της Επιτροπής και τα μέτρα που έλαβε αναφορικά με αυτή την υπόθεση είναι πολύ περισσότερο σύμφωνα με το ρόλο της Επιτροπής ως θεματοφύλακα των συνθηκών ε, σε σχέση με αυτό που έχει γίνει όσον αφορά την ελεύθερη κυκλοφορία των προσώπων. Ε, αυτό μας δείχνει ότι υπάρχει βούληση, υπάρχει τρόπος ώστε να τηρούνται οι κανόνες. Ευχαριστώ για τη σύντομη παρουσίαση. Έχουμε τον εκπρόσωπο της Επιτροπής, τον κύριο Ροντρίγκε, που θα μας πληροφορήσει για την αξιολόγηση που έχει γίνει από την Επιτροπή. Uh, good morning. Thank you. Καλημέρα και ευχαριστώ επιβεβαιώνω ότι συμφωνούμε με τον αναφέρον, τον κύριο Βάλκε. Η Επιτροπή από την αρχή κατανόησε ότι η Ισπανία είχε το δικαίωμα ε, να ζητάει πληροφορίες για περισσικά στοιχεία στο εξωτερικό. Όμως ε, βλέπαμε πάντα ότι σε περίπτωση αποτυχίας να εκπληρώσει κάποιο αυτή την υποχρέωση ήταν πολύ δυσανάλογα τα αποτελέσματα. Οι ποινέ που επιβλήθηκαν, τα πρόστιμα είναι υψηλότερα ε, σε σχέση με αυτά που αφορούν ε, εγχώριες υποθέσεις. Σε κάποιες περιπτώσεις φτάνουν στο σημείο να στερούν ε, τα περισσότερα του στοιχεία στον ιδιοκτήτη να αναγκάζεται λίγο να πουλάτε προσκευτικά για να μπορέσει να πληρώσει τα πρόστιμα. Ξεκίνησαν διαδικασίες ε, στην Επιτροπή το 2014. Στείλαμε μια επιστολή επίσημη ε, και πρόσφατα μια γνωμοδότηση και η Ισπανία συνεχίζει να επιμένει ότι δεν ε, είναι αντίθετη στην Ευρωπαϊκή Νομοθεσία η ισπανική νομοθεσία. Έχουμε επαφέ με, τις αρχέ, με διάφορες αρχές της Ισπανίας για να, κάνουμε, να έχουμε κάποια ανταλλαγή απόψεων, για να ε, δούμε πώ ε, ανταποκρίνεται στι ευρωπαϊκέ συνθήκε. Δεν ήταν επιτυχημένε οι επαφέ που κάναμε και πρόσφατα η Επιτροπή αποφάσισε στι 6 Ιουνίου του 2019 αυτό το χρόνο να παραπέμψει το θέμα στο δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τώρα είμαστε στη δικασία ε, αυτή και είμαστε σύμφωνοι απόλυτος με τον αναφέροντα και περιμένουμε την απόφαση του δικαστηρίου για να ακυρώσουμε την ε, νομοθεσία αυτή της Ισπανίας όσον αφορά το κομμάτι της αναλογίας. Είναι πολύ ενδιαφέρουσε οι πληροφορίε που μα δώσετε και σα παρακαλώ, ε, συνάδελφοι που θέλετε να πάρετε το λόγο, κύριο Φάλκε. Ε, ευχαριστώ, Πρόεδρε. Να ευχαριστήσω τον υποβάλλοντα για την αναφορά. και να σημειώσω ότι η προσπάθεια της Κομισιόν μάλλον δεν έχει εκτιμηθεί από την Ισπανική κυβέρνηση. Δηλαδή αυτή τη στιγμή περιμένουμε μία ανταπόκριση από το δικαστήριο και εμείς ε, ως μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου θα έχουμε και άλλες τέτοιες αναφορές να εξετάσουμε αν τα κράτη-μέλη συνεχίσουν με τέτοιου είδους πολιτικές. Τα πράγματα μπορεί να γίνουν ακόμη πιο σοβαρά εάν ολοκληρωθεί από αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου. Ιδιαίτερα σχετικά με ξένους υπηκόους μόνιμους κατοίκους άλλης χώρας και με τα περιουσιακά στοιχεία που κατέχουν σε άλλες χώρες. Θα πρέπει να υιοθετήσουμε λοιπόν μια νομοθεσία ώστε να προστατεύουμε τους πολίτες αυτούς. Ευχαριστούμε τον κύριο Φάλκε. Ποιος άλλος θα ήθελε να τοποθετηθεί εδώ. Δεν βλέπω εθελοντές. Λοιπόν, θα έλεγα το εξής. Να διατηρήσουμε την αναφορά αυτή ανοιχτή, να αποστείλουμε επιστολή στις Ισπανικές Αρχές, στο Υπουργείο Οικονομικών σχετικά με την αναλογικότητα των σχετικών διατάξεων, όπως και των κυρώσεων. Σχετικά με περιουσιακά στοιχεία που κατέχονται σε άλλη χώρα, των μονίμως διαμενόντων. Συμφωνούμε με το συμπέρασμα αυτό. Ωραία. Πάμε τώρα στην επόμενη αναφορά. 869 του 2018 από Ολλανδό υποβάλλοντα για τις τελευταίες εξελίξεις της έρευνας του Πλακούντα. Νόμιζα ότι θα τον είχαμε εδώ, τον Ετούντα, αλλά δεν τον έχουμε. Πάμε απευθείας λοιπόν στην απάντηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ο εκπρόσωπο, της Κομισιόν, παρακαλώ. Ε, ζητώ συγγνώμη που δυσκολεύαμε κάπω με το όνομά σα. Είστε έτοιμο. Ωραία. Έχει το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Σχετικά με την έρευνα του Πλακούντα και την ε, καταγγελία ότι δεν υπάρχουν, δεν διατίθενται επαρκή πόροι για την έρευνα αυτή. Να πω ότι λίγο ή πολύ 10 εκατομμύρια ευρώ έχουμε χρηματοδοτήσει στην έρευνα του Πλακούντα τα τελευταία πέντε χρόνια, ας πούμε, λέει ο μιλητής, σχετικά με την ατμοσφαιρική μόλυνση των ε, νεογνών και πριν τη γέννηση. Έχουν γίνει μελέτες σχετικά με την δυνατότητά μας να εξετάσουμε καλύτερα, να έχουμε καλύτερη απεικόνηση των σχετικών ιστών. να σας πω ότι δεν εστιαζόμαστε σε συγκεκριμένε νόσους ή επιστημονική περιοχή. Υποβάλλουμε ένα πλαίσιο ε, προβλήματος και από εκεί πέρα εξαιρετά από τους επιστήμονες, από τους ερευνητές. Υπάρχουν πολλά προγράμματα τα οποία όμως ε, υπακούν σε μια bottom προσέγγιση ως προς την αξιολόγησή τους. Όσο περισσότερες προτάσεις έχουμε σε μια συγκεκριμένη περιοχή, τόσο υψηλότερο προϋπολογισμό έχουμε, όπως και για, υπό το Marie Curie το πρόγραμμα. Χρειαζόμαστε λοιπόν περισσότερες υποβολές έργων και δεν βλέπουμε κάποια δυσαναλογία εμείς ή κάποια διακριτική μεταχείριση ως τα θέματα της έρευνας του Πλακούντα με ποσοστό επιτυχίας 9% είναι πάνω ή κάτω αυτό που έχουμε και με άλλες νόσους ή σε άλλες περιοχές ερεύνης ως προς τα χρηματοδοτούμενα από την Κομισιόν έργα. Κάποιο μέλος, η κυρία Κίρτον. Ευχαριστώ πρόεδρε να ευχαριστήσω την Κομισιόν για την ενημέρωση των τελευταίων πέντε ετών. Ε, πρόκειται ξεκάθαρα για μια περιοχή υψηλού ενδιαφέροντος. Τα σχόλια των υποβαλλόντων για την δυνητική συνεργασία με τις ΗΠΑ ως την έρευνα αυτή και διεθνώς για να καλύψουμε τα θέματα της ατμοσφαιρικής ρήπανσης και άλλων στοιχείων της ατμόσφαιρας, εξωγενών στοιχείων επί των βρεφών, πρέπει να ενισχυθεί, να υποστηριχθεί. Εμείς θέλουμε την αναφορά αυτή να τη διατηρήσουμε ανοιχτή και να ακούσουμε περισσότερα από την Κομισιόν σχετικά με τη διασφάλιση ε, γραμμών κονδυλίων του προπολογισμού ώστε να συνεχίσουμε να χρηματοδοτούμε τη σχετική ερεύνα. Σας ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρος. Κάποιο άλλο μέλος. Όχι εκ μέρους των Πρασίνων και εγώ υποστηρίζω ότι πρέπει να διατηρήσουμε την αναφορά ανοιχτή και να συνεχίσουμε την έρευνα. Άρα, μπορώ να θεωρήσω ότι έχουμε συμφωνήσει και σας ευχαριστώ και πολύ γρήγορα. Περνάμε στην αναφορά 204 του 2019 της ε, Evelian van den Brink, Ολλανδικής σχετικά με το αίτημα χρηματοδότησης της βιοιατρικής έρευνας για τη μυαλγική εγκεφαλομυελίτιδα. Παρουσία της αναφέρουσας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ όλους όσους τη βοήθησαν να είναι εδώ σήμερα και σας ευχαριστούμε πολύ κυρία Φάντεμπρικ που είστε εδώ και μπορούμε να μιλήσουμε μαζί σας. Να της δώσουμε το μικρόφωνο και το λόγο μαζί. Παρακαλώ, έχετε το λόγο. Δεν βιαζόμαστε, μην ανησυχείτε. Δεν είναι ανοιχτό το μικρόφωνο της δυστυχώς. nation win. Help us. President Montserrat, members of the Committee on Petitions, thank you very much for your invitation. Με πρόεδρε Μουσεράτ, μέλη τη Επιτροπή Αναφορών, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκλησή Ε, με τιμά θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Francis Martin για την εξαιρετική του βοήθεια και στήριξη, την ε, ME Action, την ben και τον, τον Ben και την ΕΣΠΕ ιδιαίτερος και τους γονείς μου. Ε, ευχαριστώ πάρα πολύ όλους όσοι στήριξαν την αναφορά μου και βοήθησαν να γίνει επιτυχία. Ε, το γεγονό ότι είμαι εδώ είναι ήδη ένα θαύμα. Για πολλά χρόνια δεν μπορούσα ούτε να μιλήσω ούτε να βγω από το κρεβάτι μου. Παρόλες τις ε, τους πολλούς περιορισμούς που έχω ακόμα και σήμερα χαίρομαι που είμαι ζωντανή, επιβίωσα. Όμως ε, δεν είναι όλοι οι ασθενείς εξίσου τυχεροί. Έχουμε χάσει πολλά εξαιρετικά μέλη της κοινότητάς μας ε, από αυτή την ασθένεια. Η ασθένεια αυτή πολύ συχνά γαλείται, αποκαλείται αόρατη και είναι αλήθεια σε κάποιο βαθμό. Χρόνιες ασθένειες μπορεί μερικές φορές να είναι αόρατες στο εξωτερικό περιβάλλον. Αλλά με την μυαλγική εγκεφαλοπάθεια αυτό είναι αλήθεια μόνο σε ένα βαθμό και γίνεται πολύ ορατή κάποια στιγμή. Ε, και μάλιστα περιγράφεται ως ζών θάνατος, ζωντανός θάνατος. Αυτός είναι ο Whitney Dafoe ο γιος του, της Janet Dafoe και του Roland Davis, καθηγητή της βιοχημίας και γενετικής στο Πανεπιστήμιο του Στάνφορντ, πολύ γνωστός ε, διάσημος επιστήμονας ε, που είχε συμμετάσχει και στο ε, σχέδιο για το ανθρώπινο γονιδίωμα, το Human Genome Project. Εργάζεται άοκνα για να θεραπεύσει το, την, το γιο του. Αυτή, ήταν η, αυτή είναι η Έλισον Hunter, ήταν ένας πολύ ζωντανό κορίτσι γεμάτο ζωή. Πέθανε στα 14 της εξαιτίας ε, της αυτή ε, και επιπλοκών προέκυψαν από αυτήν. Αυτό είναι ο Μάρκ Βίνκ. Ήταν γιατρός και έτρεχε το μαραθώνιο. Τώρα Ακόμα και να περπατήσει μέχρι την ε, τουαλέτα είναι πολύ πιο δύσκολο οποιοδήποτε μαραθώνιο είχε τρέξει. Και αυτή είμαι εγώ, σε μία από τις χειρότερες στιγμές μου. Ε, είμαι ασθενό εδώ και πάνω από 20 χρόνια. Και εδώ είμαι εγώ ως παιδί. Ε, θυμάμαι με πολύ χαρά την ζωή μου όταν ήμουν υγιής. Μια φορά μάλιστα είχα καταφέρει να ε, καβαλήσω και ένα άλογο χωρίς σέλα. Ε, η ασθένεια αυτή είναι αόρατη μόνο, σε αυτό το βαθμό μόνο όταν οι, οι άνθρωποι προτιμούν να κοιτάξουν προς άλλη μεριά. Ε, και αυτό είναι αυτό που συμβαίνει, γιατί οι ασθενείς ε, ε, υποφέρουν από την σιωπή. το γεγονός ότι δεν είναι πολύ γνωστά τα αίτια και δεν υπάρχει διαγνωστικό τεστ έχει δημιουργήσει ένα τρομακτικό στίγμα. πολλοί μας λένε είναι στο κεφάλι σου η ασθένεια και πολύ συχνά δεν παίρνουμε την κατάλληλη θεραπεία γιατί ακριβώς υπάρχει λαθασμένη εικόνα για την ασθένεια και ανεπαρκής ε, συγγνώμη, ε, επιστημονική πρόοδος. Ο, παλιά τον καρκίνο, ε, για τον καρκίνο έλεγαν ότι προκύπτει από την καταπίεση κακών σκέψεων, ότι η δική μας ασθένεια ήταν ιστερική παράλυση και το AIDS ήταν εξαιτία του στρες που να είναι κανείς ομοφιλόφιλος. Ευτυχώς έχουν αλλάξει οι καιροί και τώρα πια ε, η αλλαγή αυτή έχει γίνει ε, χάρη στην επιστήμη, όχι χάρη στη σιωπή. Γι' αυτό είμαι εδώ σήμερα. Χρειάζεται περισσότερη χρηματοδότηση στην βιοιατρική έρευνα για την ε, μυαλική εγκεφαλομυελίτιδα. Πρέπει να, είμαστε, να έχουμε ένα ικανό διαγνωστικό ε, τεστ και ε, να λαμβάνουμε την κατάλληλη θεραπεία. Οι επιστήμονες έχουν κάνει σημαντική πρόοδο με ιδιωτικά κεφάλαια αλλά και με δημόσια και κρατικά κεφάλαια στις ΗΠΑ από το NIH. Ε, τα, πιο μεγάλα αμερικανικά πανεπιστήμια έχουν ειδικά ερευνητικά προγράμματα για αυτή την ασθένεια. Ε, και έχουμε ήδη σημαντική πρόοδο. Είμαι πεπισμένη ότι ως Ευρωπαίοι μπορούμε να, κάνουμε πολύ περισσότερα για να λύσουμε το πρόβλημα αυτής ε, της ε, ασθένειας την οποία έχουμε αμελήσει το για τόσο καιρό. Έχουμε εξαιρετικούς επιστήμονες αλλά που θέλουν με ενθουσιασμό να δουλέψουν αλλά χρειάζονται χρηματοδότηση και χρειάζεται μια μακρόχρονη δέσμευση με ισότιμη χρηματοδότηση και μια συνολική στρατηγική. Δεν είναι μόνο ε, ανθρωπιστικό ή ηθικό το ζήτημα. Αν οι ασθενείς γυρίσουν στην δουλειά τους, θα υπάρχουν και οικονομικά ωφέλη για την συνολική οικονομία. Εγώ πιστεύω στην Ευρώπη και στις κοινέ μας αρχές της ισότητας, της δικαιοσύνης ε, και των ίσων ευκαιριών. Είμαι απολύτως ε, πεπισμένη ότι μπορούμε ουσιαστικά να βοηθήσουμε για να λυθεί το πρόβλημα αν το προσπαθήσουμε. Εκ μέρους όλων των ασθενών σας ζητώ παρακαλώ πολύ μη γυρνάτε το βλέμμα σας αλλού. Είμαστε εδώ και είμαστε ορατοί. Παρακαλώ πολύ βοηθήστε μας να γυρίσουμε στην κανονική μας καθημερινή μας ζωή. Ε, με, την, ε, με ελπίδα και αποφασιστικότητα μπορούμε να λύσουμε το πρόβλημα μαζί. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε. Ε, Ευέλιαν. Πραγματικά έκανες ε, το πρόβλημα αυτό ορατό. Ε, θα δώσουμε το λόγο σε έναν εκπρόσωπο της ε, Κομισιόν. Στον εκπρόσωπο της Κομισιόν. Ευχαριστούμε πολύ την κυρία Φάντεν Μπρίνκ για αυτή την μαρτυρία της. Δυστυχώ, ε, θα παραλάβω αυτό που είπα πριν, δεν έχουμε προγράμματα για συγκεκριμένε ασθένειε εμεί στην Κομισιόν. Δεν εστιάζουμε σε συγκεκριμένε ασθένειε. Έχουμε ε, προκηρύξουμε ε, την διαδικασία συμμετοχής και οι ίδιοι επιστήμονες μας υποβάλλουν προγράμματα. Ε, την περασμένη εβδομάδα, για παράδειγμα, είχαμε μια πρόταση για μια καινούργια παρέμβαση για τι χρόνιες ασθένειε. Εκεί θα μπορούσε να γίνει έρευνα και για αυτή την ασθένεια. Ίσως ε, δεν κάνουμε αρκετά έτσι ώστε να παροτρύνουμε τους ε, επιστήμονες να υποβάλουν περισσότερες προτάσεις και να δουλέψουν περισσότερο. Οι, οι μικρές εισαγωγικά ασθένειες ε, λέγεται ότι δεν αξιολογούνται τόσο πολύ όσο οι μεγάλες ασθένειες. Έτσι λέγεται, αλλά εμείς όταν κάνουμε την αξιολόγηση των προτάσεων λέμε ότι το σημαντικό είναι οι, οι συνέπειες που θα έχει η έρευνα εντός της κοινότητας των ασθενών, όχι συνολικά σε όλο το φάσμα των ασθενών. Οπότε δεν υπάρχουν άλλα κριτήρια για τις μικρές και άλλα για τις μεγάλες. Οπότε η απάντησή μου είναι ότι θα πρέπει να βρούμε τρόπους να παροτρύνουμε ακόμη περισσότερο τους επιστήμονες να συμμετάσχουν. Ε, ο, Είχαμε πολύ μικρό ποσοστό επιτυχίας στο, στην αρχή του ορίζον 2020, 2-3%, αλλά στο τέλος του ορίζον 2020 το ποσοστό αυτό έχει αυξηθεί γύρω στο 20%, οπότε θα έχουμε περισσότερες ευκαιρίες, ελπίζω. Η σύγκριση με το NIH, στο οποίο αναφερθήκατε, ε, των Ηνωμένων Πολιτειών, ναι, πραγματικά κάνουν πολλά, αλλά έχουν και έναν προπολογισμό 30 φορές πιο πολύ από τον προπολογισμό της Κομισιόν. Αυτοί έχουν 30 δισεκατομμύρια το χρόνο, εμείς είμαστε περίπου στο 1 δισεκατομμύριο το χρόνο. Οπότε έχουν πολύ περισσότερα μέσα. Επίσης το 95% των, της κρατικής χρηματοδότησης στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι, προέρχεται από τα κράτη-μέλη και μόνο το 5% από την Κομισιόν. Οπότε πρέπει να πιέσετε και τις εθνικές αρχές για να αφιερώσουν μεγαλύτερα κονδύλια. Thanks. Uh, very... Πρόεδρος, ευχαριστούμε πολύ. Ποιος θέλει το λόγο? Ποιος Πάλμερ. Να ευχαριστήσω την αναφέρουσα για τη μαρτυρία της δεν κάνετε απλά ορατού του ασθενεί με μελική εγκεφάλο, αλλά είστε η φωνή του στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και πιστεύω ότι θα είναι περήφανοι για αυτή τη συνεισφορά σα σήμερα το πρωί. Θέλω να σα ευχαριστήσω λοιπόν και όλους όσους υποστήριξαν αυτή την αναφορά, ακόμα και την δικιά μου εκλογική περιφέρεια που υποστηρίζει τους ασθενείς εδώ και πάρα πολλά χρόνια με προσωπικές θυσίες. Συναντήθηκα με την Διεθνή ε, Συμμαχία για την μυαλγική κεφαλομυελίδα, η οποία χρειάζεται περισσότερη επιστημονική έρευνα. Όπως αναφέρθηκε πριν, είναι μια πάθηση που αφορά 20 εκατομμύρια ανθρώπους σε όλο τον κόσμο. Είναι μια καταστροφική για αυτούς ε, νόσος. Και όπως ε, είπε και η αναφέρουσα, θα πρέπει να δούμε το θέμα σοβαρά και να ηγηθούμε τις προσπάθειες του ιατρικού κλάδου ε, σε παγκόσμιο επίπεδο. Το κόστος είναι πολύ μεγάλο και το οικονομικό αλλά και το κόστος ε, στα άτομα, στους φροντιστές τους και τις οικογένειές τους. Σήμερα το πρωί λοιπόν, αυτή τη στιγμή θέλω να υποστηρίξω αυτό που είπανε πάρα πολύ από τους ψηφοφόρους μου και να πω στην Επιτροπή ότι πρέπει να βρεθεί η κατάλληλη χρηματοδότηση για να υπάρξει αυτή η βιοετρική ε, έρευνα, διαγνωστικά τεστ που θα είναι αξιόπιστα για την μυαλική κεφαλαιομελίτιδα αλλά και έρευνα για την θεραπεία ζητά από την Επιτροπή να είναι πιο συγκεκριμένη. Απλά να ε, βρει την κατάλληλη χρηματοδότηση γιατί είναι μία νόσος, είπε πολλές φορές δεν, ε, στην οποία δεν γίνεται η διάγνωση. Υπάρχει μια παρεξήγηση λοιπόν, γιατί δεν γίνεται πολλές φορές σωστή διάγνωση και υπάρχουν ε, διάφορα, διάφορες προκαταλήψεις σχετικά με τους ανθρώπους που πάσχουν από αυτή την ε, πάθηση. Στην ακρόαση ε, του υποψήφιου τρόπου για την υγεία είδα ότι ήταν πολύ φιλόδοξος για την ατζέντα στο θέμα της ε, υγείας. Υπάρχει ε, ομοφωνία, συνένεση στα όργανα ότι θα πρέπει να στηριχθεί η βιοτρική έρευνα για τη διάγνωση και τη θεραπεία της μελικής εγκεφαλομιελίτιδης. Θα ήθελα Επομένω, να μην ανοιχτεί αυτή η αναφορά για να μπορέσουμε να παρακολουθήσουμε την κατάσταση και το έργο της Επιτροπής και ενδεχομένω σε κάποιους μήνες θα μπορούμε να έχουμε μία πιο ελκυστική, ε, πιο ενδιαφέρουσα ιστορία, να διηγηθούμε για το θέμα αυτό και να διορθώσουμε την μεγάλη αδικία για την υποχρηματοδότηση της έρευνας για την μυαλγική εφαλομιλίτιδα σε σχέση με τις άλλες ασθένειες και νόσους. Ευχαριστώ κύριε Πάλμερ. Ο κύριος Μπούσμαν. Παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ. Και στην κυρία Φαντεμπρίνγκ που ήταν εδώ σήμερα και που μας παρουσίασε την κατάσταση. Ευχαριστώ και την βοηθό που την διευκόλυνε. Ασχολήθηκα με την νόσο αυτή και είναι μια πολυστημική ε, χρόνια πάθηση που επηρεάζει δραστικά τη ζωή των ασθενών. Η Ο βασικός λόγος, η αιτία της ασθένειας είναι άγνωστη, από όσο γνωρίζω. Ε, μιλάμε για μια κατάσταση χρόνιας κόπος που μπορεί να κρατήσει έξι μήνες αδυναμίας. Είναι παθολογικό το όριο της εξάντλησης και είναι πολύ υψηλή επιβάρυνση που αισθάνονται οι ασθενείς. Ο ύπνος επίσης δεν βοηθάει, δεν βοηθάει στην ξεκούραση και υπάρχουν και άλλα συμπτώματα που μοιάζουν με τη γρήπη, που έχουν να κάνουν με πόνο στους μυς, στα άκρα, φλεγμονές κτλ. Αυτό σημαίνει φυσικά για τους ασθενείς πολύ χαμηλό, χαμηλή ποιότητα ζωής. 60 με 80% δεν είναι ικανοί να εργαστούν, και κάποιοι ε, χρήσουν ιδιαίτερης ε, φροντίδας. Εδώ και δύο μέρες αναγνωρίστηκε αυτή η ασθένεια στην ε, Ολλανδία. Ε, ψηφίστηκε ε, αυτή η απόφαση στην, τον Οκτώβριο. Επίσης υποστηρίζεται η χρηματοδότηση έρευνας αυτής στη συνέχεια και γι' αυτό θα ήθελα να παραμείνει ανοιχτή η αναφορά. Muchísimas gracias. Ευχαριστούμε. Για να ολοκληρώσουμε το σημείο έχετε πάλι δύο λεπτά ή υποβάλλουσα, παρακαλώ. I would Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους ε, για την στήριξή σας. Πολύ χαίρομαι που εισακούστηκα, που με ακούτε, ότι αντιλαμβάνεστε δηλαδή ότι η ανάγκη για μια αλλαγή εδώ είναι πραγματική και επίγουσα πρέπει αυτές οι αλλαγές να λάβουν χώρα και ε, αυτή η ελπίδα να μετατραπεί σε ανάληψη δράσης, σε πράξη δηλαδή που θα βελτιώσει τη ζωή διαφορών ανθρώπων. Σας ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστούμε πολύ που ήσασταν εδώ μαζί μας. Πραγματικά θα κάνουμε ό,τι μπορούμε σχετικά με την συνέχεια που θα δοθεί στην αναφορά αυτή, έχοντας ακούσει και την Κομισιόν και τις πολιτικές ομάδες. Θα διατηρήσουμε ανοιχτή την αναφορά σας αυτή για να συνεχίσουμε να συνεργαζόμαστε στο θέμα αυτό και θα ζητήσουμε τη διευκόλυνση της ενημέρωσής μας σχετικά με την επικαιροποίηση που θα έχουμε για τα όσα αντιμετωπίζετε και εσείς και οι υπόλοιποι που αντιμετωπίζουν την όσα αυτή. Έχουμε πολλά να πούμε και για τα κονδύλια τα αφιερωμένα στην έρευνα. Δεν πρόκειται να εγκαταλείψουμε το θέμα. Θα συνεχίσουμε να δουλεύουμε από κοινού μαζί με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή τις πολιτικές ομάδες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για να υποστηρίζουμε διαρκώς την έρευνα, για να διατηρήσουμε ανοιχτή την αναφορά σας και να μπορέσουμε πραγματικά να σας βοηθήσουμε. Σας ευχαριστώ πραγματικά θερμότατα για την παρουσία σας. Μας βοηθάτε. Ευχαριστώ. Al último Πάμε τώρα στην τελευταία αναφορά 371-2018 εκ μέρους της ΑΠΙΚΟ για την ε, κοινωνική ενσωμάτωση ε, παιδιών που, με αναπηρία όπως και την 2582 του 2013 του κυρίου Διαλόνθο Αλόνσο Παθ για τις διακρίσεις που υφίστανται παιδιά με ειδικές ανάγκες ή αναπηρία από τις Ισπανικές αρχές. Δεν βρίσκονται οι αναφέροντες στην αίθουσα, αλλά μας ε, παρακολουθούν με βίντεο link ε, και έχουν και μήνυμα το οποίο θα σας ε, μεταβιβάσουμε αυτή τη στιγμή. Καλημέρα στα μέλη της ε, Επιτροπής Αναφορών. Το 2015 είχαμε λάβει απαντήσεις ε, στην αναφορά μας που απευθυνόταν προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ώστε στα πλαίσια των άρθρων 20, 21, 24 και 26 της Χάρτας των και Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης να εξεταστεί η περίπτωση των διακρίσεων ε, του 2013 ενός από τους γιους μου που είχε απορριφθεί από, Ισπανία, από σχολείο στην Ισπανία ε, λόγω της αναπηρίας του. Η Επιτροπή είχε καταλήξει στο συμπέρασμα ότι η περίπτωση αυτή δεν ενέπιπτε στην αρμοδιότητα των ε, θεμάτων υπό το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτή τη στιγμή μετά από ε, την παρακολούθηση στον στο Σαν Κριστόβαλ της ε, Λαλαγούνα σε κανονικό σχολείο ε, μαθαίνω ε, με έκπληξη ότι η Επιτροπή αποφάσισε να επανεξετάσει το θέμα και αποφάσισε ότι εμπίπτει στην αρμοδιότητά της πολλά, με τα χρόνια που έχουν περάσει ε, όχι μόνο με τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε από την απόρριψη αλλά και επειδή θεωρώ ότι είναι καθήκον των εκπροσώπων μας ε, στη, στα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα να αντιμετωπίζουν τα θέματα ε, διάκρισης ε, και κοινωνικού αποκλεισμού των ανθρώπων που αντιμετωπίζουν προβλήματα αναπηρίας. Στο εκπαιδευτικό σύστημα στην Ισπανία δεν αναγνωρίζονται τα δικαιώματα συμμετοχής όλων ιδιαίτερα υπό το άρθρο 24 της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των ανθρώπων που αντιμετωπίζουν αναπηρίες, η οποία έχει ενσωματωθεί ως διάταξη στο Ισπανικό Δίκαιο το 2008. Και παρά την έκθεση των Ηνωμένων Αθνών του 2017 σχετικά με το, ε, ε, πρότυπο το εκπαιδευτικό της Ισπανίας που ακολουθεί διακριτική μεταχείριση σε κάποιες περιπτώσεις. Έχουμε την νομοθεσία, στην παιδεία, ε, την νομοθεσία για την ε, παιδεία στην Ισπανία από το 2006 και το 2013 σχετικά με τα εκπαιδευτικά κέντρα που πρέπει να τηρούν συγκεκριμένα χαρακτηριστικά για παιδιά όλων των ηλικιών που αντιμετωπίζουν συγκεκριμένες εκπαιδευτικές ανάγκες οι οποίες ανάγκες ε, ε, αποκλίνουν ε, με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά από τον μέσο όρο. Είναι αναγκαιότητα να αναγνωρίσουμε τις ανάγκες της διαφορετικότητας και η κοινωνία εν γέννη να αναγνωρίζει τις ιδιαίτερες ανάγκες και τα χαρακτηριστικά των παιδιών αυτών. Να μην να μην ασκούνται διακρίσεις κατά των παιδιών όπως το δικό μου, και θα πρέπει ε, να μπορούμε να βλέπουμε τα παιδιά αυτά ως μέλη της κοινωνίας και να μην απομακρύνονται, να μην στιγματίζονται, να μην επικρατούν ε, στερεότυπα στην κοινωνία σχετικά με το πρόβλημά τους. Επομένως δεν κατανοώ παρά την επέκταση της οδηγίας 78 ε, του 2000 του Συμβουλίου που απαγορεύει τις διακρίσεις ε, ε, λόγω αναπηρίας, ηλικίας, ε, σεξουαλικής προτίμησης, η περίπτωση των παιδιών όπως του γιού μου είναι μια περίπτωση που αποκλίνει από, τις, από την χρηστή εφαρμογή των διατάξεων του δικαίου Ιδιαίτερα για άτομα, για παιδιά δηλαδή, που είναι, ε, δεν είναι σε θέση να υπερασπιστούν πλήρως τα δικαιώματά τους ατομικά. ελπίζω πραγματικά η αναφορά αυτή, το πρόβλημα αυτό, να έχει κρούσει τον κόδωνα του κινδύνου σχετικά με όλα τα άτομα που αντιμετωπίζουν τέτοια προβλήματα σε οποιαδήποτε χώρα, σε οποιαδήποτε περιφέρεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ώστε να εφαρμόζονται οι διατάξεις ε, για τα ανθρώπινα δικαιώματα των πιο ευάλωτων μελών της κοινωνίας. Γιατί έχουμε φαινόμενα κοινωνικού αποκλεισμού, απομόνωσης ε, για τους ανθρώπους που αντιμετωπίζουν τέτοια προβλήματα αναπηρίας. Θα ζητούσα λοιπόν από την Επιτροπή σας να ενεργοποιήσει τον, τους απαραίτητους μηχανισμούς ώστε όλες οι περιφέρειες της ε, Ένωσης να αποκλείουν αυτές τις, αυτή τη διακριτική μεταχείριση και να εφαρμόζουν μια ε, εκπαιδευτική πολιτική για την καλύτερη κατανόηση της διαφορετικότητας που να εντάσσεται στον 21ο αιώνα στην ενημέρωση που έχουμε σήμερα ως προς την διαφορετικότητα και την αξία που έχουν όλα τα μέλη της κοινωνίας. Νομίζω λοιπόν ότι όλοι αξίζουμε μια ε, ποιοτική παιδεία και εδώ δεν, καθόλου δεν αξιώνω την αποζημίωση των προβλημάτων που αντιμετωπίσαμε όλα τα χρόνια, αλλά την αποκατάσταση. Σας ευχαριστώ, λέει η Πρόεδρος. Ο κύριος Σομπτερέκε, όχι, η κυρία Πορέρο πρώτα. Buenos días. Καλή σας μέρα. Θα πω δύο λόγια στα ισπανικά, μια και ο αναφέρον μίλησε στα ισπανικά. Είχαμε πάρει το κείμενο του και γραπτά, αλλά είναι άλλη αίσθηση που δημιουργείται όταν ακούμε αυτό τον πατέρα να μιλάει μέσω του βίντεο και θα ήθελα να πω ότι πραγματικά συμμερίζομαι καταρχήν την ε, κατάσταση στην οποία βρίσκεται. Προφανώς δεν είναι ο μόνος, δυστυχώς. Η Κομισιόν στο πλαίσιο των δυνατοτήτων της προσπαθεί να κάνει ό,τι μπορεί για να προχωρήσουμε στην Ευρώπη σε μια εκπαίδευση που δεν θα αφήνει κανέναν εκτός, που θα είναι ποιοτική για όλα τα άτομα με αναπηρίες. Στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων μας βέβαια. Και τώρα θα περάσω στα αγγλικά, αν μου επιτρέπετε. Να σας πω μερικές, να σας δώσω μερικές λεπτομέρειες για το έργο μας. Με πολύ ενδιαφέρον και πραγματική ανησυχία Διαβάσαμε τις ε, περαιτέρω πληροφορίες που έστειλε ο αναφέρον και τη γνώμη και των άλλων οργανώσεων. Δυστυχώς η κατάσταση δεν έχει αλλάξει. Οι αρμοδιότητες ε, στον τομέα της εκπαίδευσης ε, πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας είναι, είναι εθνικές. Παρ' όλα αυτά στο μέτρο που μας επιτρέπουν οι αρμοδιότητές μας, εμπνεόμενοι από την Ευρωπαϊκή Σύμβαση για τα Δικαιώματα των ανθρώπων με Αναπηρίες, ε, προσπαθούμε να λάβουμε δράση. Η σύμβαση είναι πάρα πολύ σαφής. Δικαίωμα στην εκπαίδευση για όλα τα άτομα αναπηρίες, χωρίς διακρίσεις, με ίσες ευκαιρίες και όχι οποιαδήποτε εκπαίδευση, αλλά εκπαίδευση ποιοτική, παροχή στέγης, ε, εξατομικευμένα μέτρα και επαρκώς ε, ενημερωμένους ε, και εκπαιδευμένους δασκάλους και καθηγητές. Οπότε εμείς στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων μας τι μπορούμε να κάνουμε, συνειδητοποίηση, να βοηθήσουμε στη συνειδητοποίηση, προάγουμε την εκπαίδευση χωρίς διακρίσεις και εξαιρέσεις, Έχουμε μια ομάδα υψηλού επίπεδου για τις αναπηρίες και συμμετέχουμε σε διασκέψεις όπως η Ευρωπαϊκή μέρα για άτομα με αναπηρία. Εκεί στηρίζουμε ε, την υπηρεσία για την, την ε, υπηρεσία για την ε, εκπαίδευση χωρίς εξαιρέσεις και πλέον και επιπλέον στην πρότασή μας για την προστασία από τις διακρίσεις, ε, μεταξύ άλλων έχουμε συμπεριλάβει και τα άτομα με αναπηρίες και τον τομέα της εκπαίδευσης. Αυτή είναι μια εκθέση του 2008 και η επιλεγμένη, η ορισμένη ως Επίτροπος κυρία Ντάλη, ε, εδώ σε αυτή τέσσερις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ανέφερε το τι μπορεί να κάνει, τι μπορούμε να κάνουμε ως Κομισιόν, ανέφερε ότι είναι αποφασισμένη να καταπολεμήσει τις διακρίσεις. Να σα πενθυμίσω επίσης ότι η Ισπανία έχει, είναι ε, συμβαλόμενο μέρος τη ε, Ευρωπαϊκή Σύμβασης για τα Δικαιώματα των Ατόμων Αναπηρία και υπάρχει δυνατότητα να χρησιμοποιηθεί και το νομικό πλαίσιο της σύμβασης για να επιτευχθεί πρόοδος στην Ισπανία. Ας το έχει αυτό υπόψη του ο ε, αναφέρον. Ευχαριστώ πολύ. Muchas gracias. Πρόεδρος, κύριε Σαλίβα. Ευχαριστώ πολύ τον αναφέροντα που θίγει αυτό το σημαντικό θέμα. Η εκπαίδευση χωρίς εξαιρέσεις, χωρίς αποκλεισμούς είναι απόλυτα σημαντικό στοιχείο για τους ανθρώπους με αναπηρία ε, θα πρέπει να αναπτύξουν τα προσόντα τους, ε, τις δεξιότητές τους έτσι ώστε να συμμετάσχουν πλήρως στην κοινωνία. Όλα ξεκινούν από την εκπαίδευση. Οπότε το τα εκπαιδευτικά μας συστήματα θα πρέπει να έχουν μαθητές ε, όλων των τύπων και να δίνουν στα άτομα με αναπηρίες τις δυνατότητες και τα μέσα έτσι ώστε να αντιμετωπίσουν τους τους με ίσες ευκαιρίες. Δεύτερον, συμφωνώ με τις παρατηρήσεις τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Άτομα, παιδιά με αναπηρίες θα πρέπει να εντάσσονται στο γενικό εκπαιδευτικό σύστημα και να τους χορηγείται επαρκής συνδρομή. Αυτό αναφέρεται και στην σύμβαση του ΟΗΕ για τα δικαιώματα των ανθρώπων με αναπηρίες, των ατόμων με αναπηρίες, που αναφέρει πως τα παιδιά με αναπηρίες πρέπει να χαίρουν ίσων ευκαιριών στην εκπαίδευσή τους. Όπως είπε η Κομισιόν, η Ισπανία όχι μόνο είναι συμβαλλόμενο μέρος της σύμβασης αυτής, αλλά έχει επίσης επικυρώσει και το ε, πρωτόκολλο ε, της σύμβασης αυτής. Παρ' όλα αυτά, εκατομμύρια παιδιά έχουν εξαιρεθεί ε, από το Γενικό Σύστημα Εκπαίδευσης ε, στην Ισπανία και αυτό θα πρέπει να ερευνηθεί. Θα πρέπει να στείλουμε επιστολή στις Ισπανικές Αρχές για το ζήτημα αυτό. Δεν θα πρέπει να γίνονται διακρίσεις, θα πρέπει τα παιδιά με αναπηρίες να εντάσσονται πλήρως στο εκπαιδευτικό σύστημα. Gracias. Πρόεδρος, ευχαριστώ. Θέλει κανείς άλλο το λόγο. Κύριε Σπουρόρη. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Για την αναφορά αυτή που υπέβαλε ένας συμπολίτης μας, ιδιαίτερα για διακρίσεις κατά παιδιών, δεν μπορεί αυτές οι διακρίσεις ε, να υπερβαίνουν το δικαίωμά τους στην παιδεία που είναι αναφέρεται το δικαίωμά τους ε, η περίπτωση των οκτώ αυτών παιδιών ε, με αναπηρία στην Ισπανία δείχνουν τα προβλήματα που έχουμε στην, ε, στον τομέα της εκπαίδευσης και στα δικαιώματά τους τα οποία δεν ε, είμαστε σε θέση να εγγυηθούμε από ό,τι φαίνεται. Μιλούμε για τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών σχετικά με τους ανθρώπους με αναπηρίες για την προστασία των δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ανθρωπίνων δικαιωμάτων, δηλαδή των ανθρώπων με αναπηρίες και ζητώ από τις Ισπανικές αρχές να εξασφαλίσουν, μάλλον να εφαρμόσουν την, ε, να προστατεύσουν τα δικαιώματα των παιδιών αυτών, των ανθρώπων αυτών, όχι μόνο ως προς διατάξεις του δικαίου που έχουμε, αλλά και στο άγραφο δίκαιο για την ε, σωστή ενσωμάτωση στην κοινωνία, για τη σωστή συμμετοχή των παιδιών αυτών. Αλλά και για τη στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, για, τις, ε, για τους ανθρώπους με αναπηρία, για τη διαφορετικότητα και για το σεβασμό των δικαιωμάτων και των οικογενειών τους. Σας ευχαριστώ. Ο κύριος Κώσα. Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε. Εκ μέρου του ΕΛΚ ε, συμφωνώ απολύτως με τους συναδέλφου που μίλησαν πριν από μένα. Αναφέρθηκαν σε κάποια στοιχεία που δεν θα ήθελα να επαναλάβω. Προφανώς ε, και ε, ο χάρτης θεμελιωδών δικαιωμάτων είναι εδώ ένα βασικό πλαίσιο, το άρθρο 24 της Σύμβασης αναφέρει ρητά ότι τα παιδιά με αναπηρίες δεν μπορούν να αποκλείονται από τα ε, τακτικά προγράμματα εκπαίδευσης. Επομένως το 24.2 είναι η πολύ βασική διάταξη εδώ. Η σύμβαση χρησιμοποιεί ευέλικτη διατύπωση γενικώ, αλλά στα θέματα παιδείας είναι προφανές ότι τα παιδιά που αντιμετωπίζουν αναπηρίες δεν μπορούν να αποκλείονται από τα εκπαιδευτικά προγράμματα. Πρέπει λοιπόν να προστατεύσουμε τα δικαιώμά τους και πρέπει να ζητήσουμε από τις Ισπανικές αρχές λεπτομερή έκθεση σχετικά με τα μέτρα που σκοπεύουν να αναλάβουν στο μέλλον προκειμένου να εξασφαλίσουν ότι δεν θα υπάρξει ξανά αποκλεισμό ε, των παιδιών από το δικαίωμά του στην παιδεία. Όπως ανέφεραν οι συνάδελφοι, η Ισπανία είχε υπογράψει και το εθελοντικό πρωτόκολλο, το οποίο προβλέπει τη σύμβαση, που προβλέπει ότι τα ενδιαφερόμενα μέρη μπορούν να προσφύγουν στα Ηνωμένα Έθνη. Και εδώ είναι μια σημαντική ευκαιρία να εμπλακούν και οι φορεί των Ηνωμένων Εθνών στην περίπτωση αυτή την Ισπανική. Και ίσως και άλλα κράτη-μέλη στην Ευρωπαϊκή Ένωση να αντιληφθούν πόσο σημαντική είναι η παιδεία. Εγώ προτείνω να συνεχίσουμε να εξετάζουμε το θέμα και να το παρακολουθούμε. Σα ευχαριστώ πολύ, λέει ο Πρόεδρος. Αν συμφωνείτε, θα πω και εγώ δύο λόγια, όχι ω πρόεδρο, αλλά ω μέλο τη επιτροπή ήμουν υπουργό υγεία ε, και κοινωνική ασφάλιση ε, στην ε, Ισπανία. Είμαστε υπερήφανοι που είχαμε υπογράψει τη σύμβαση και όλα τα πρωτόκολλα. Μαζί με την οργάνωση Θέρμη στην Ισπανία για την υποστήριξη των ανθρώπων με αναπηρίες. Ήθελα να σας πω το εξής. Στην Ισπανία έχουμε ένα 83% ενσωμάτωσης στα τακτικά σχολεία των ανθρώπων με αναπηρίες. Οι γονείς εκείνοι που αποφασίζουν να συνεχίσουν σε κέντρα εξειδικευμένα, καλώς. Όσοι όμως αποφασίζουν στα κανονικά σχολεία να συνεχίσουν τη μόρφωση των παιδιών τους, έχουμε εκεί αυτό το ποσοστό απορρόφησης, αν θέλετε, ενσωμάτωση 83%. Υπάρχουν άλλα κράτη-μέλη, ε, έχουμε πολύ διαφορετικά συστήματα εκπαιδευτικά, αλλά αν δούμε περίπου τον μέσο όρο, δεν ξεπερνούμε το 50% κατά πολύ ε, στην ενσωμάτωση. Επομένως η Ισπανία έχει καταβάλει σημαντικές προσπάθειες να ενσωματώσει τα παιδιά αυτά που αντιμετωπίζουν αναπηρίες για την ενσωμάτωσή τους, την παρακολούθηση των τακτικών προγραμμάτων εκπαίδευσης στα σχολεία. Εγώ λοιπόν προτείνω να διατηρήσουμε ανοιχτή την αναφορά αυτή. Η προσωπική μου πρόταση ως μέλος είναι να αποστείλουμε επιστολή στις Ισπανικές αρχές και στις περιφερειακές αρχές της Ισπανίας ώστε να μας εξηγήσουν για ποιον λόγο δεν μπόρεσαν αυτά τα παιδιά να παρακολουθήσουν τα κανονικά προγράμματα εκπαίδευσης και πραγματικά θα συνέστηνα θερμά στον ε, αναφέροντα ε, μαζί με άλλες οργανώσεις που έχουμε στο έδαφος στην Ισπανία, μαζί με τη Θέρμη, η οποία συνεργάζεται ε, με διάφορους κυβερνητικούς φορείς στην Ισπανία. Νομίζω ότι πραγματικά στη χώρα μας προσπαθούμε να υποστηρίξουμε και τη διαφορετικότητα και τους ανθρώπους με αναπηρία και έχουμε ένα από τα υψηλότερα ποσοστά ενσωμάτωσης όπως σας έλεγα. Τώρα η Επιτροπή μας ζήτησε να τοποθετηθεί και αυτή, ιδιαίτερα για την 371 αναφορά, ε, ο κύριος Σοπντεμπέκε. Παρακαλώ. Ε, good morning everybody. Καλημέρα. Να κάποια πράγματα παραπάνω για αυτή την αναφορά. Δώσουμε την απάντησή μας και στη συγκεκριμένη περίπτωση οι αρμοδιότητες αναπόκειται στα κράτη-μέλη. Ξαναβλέποντας το θέμα, ίσως κάτι έχουμε παραλύσει γιατί κάτι που είναι πολύ σημαντικό για την υπόθεση αυτή είναι ότι 8 με αυτές που αρνήθηκαν ε, είσοδο σε σχολή επαγγελματική ε, κατάρτιση είναι μια λεπτομέρεια σημαντική γιατί η επαγγελματική εκπαίδευση καλύπτεται από την οδηγία ε, ε, για την ισότητα στην ε, εργασία και καλύπτει και την επαγγελματική κατάρτιση. Επομένω, με βάση αυτή την οδηγία θα μπορούσαμε να πούμε ότι θα μπορούσε να γίνει προσφυγή στο Ισπανικό Δικαστήριο γιατί έχουμε διάκριση με βάση την οδηγία του ε, για την ε, ισότητα στην ε, απασχόληση. Αποκλείστηκαν αυτοί με αυτές από ένα σχολείο επαγγελματική κατάρτισης και αυτό δεν βοηθάει πολύ για την καταπολέμηση της μια αποδοχή από άλλα σχολεία γενική εκπαίδευση. Αυτό το σημείο θέλω να προσθέσω στα αυτά που προϋπόθηκαν. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστούμε και εμείς, λέει η Πρόεδρος. Και ως μέλος και ως Πρόεδρος προσπαθώ να είμαι όσο πιο αντικειμενική μπορώ. Και αν συμφωνείτε, καθότι αυτό μου διαβίβασαν και οι εκπρόσωποι των πολιτικών ομάδων, λέω να διατηρήσουμε ανοιχτή την αναφορά. Αν κάποιο έχει αντίρρηση παρακαλώ να μου το πει. Γιατί σας είπα, προηγουμένω τοποθετήθηκα ως μέλος και όχι ως πρόεδρος. Προτείνω λοιπόν να διατηρήσουμε ανοιχτή την αναφορά, να αποστείλουμε επιστολή στις ε, Ισπανικές αρχές, στο αρμόδιο Υπουργείο και άλλους φορεί, ώστε οι, οι Ισπανικές αρχές να υποστηρίζουν τις ανάγκες των παιδιών και των ανθρώπων με αναπηρίες. Να συστήσουμε, να προτείνουμε στον αναφέροντα να έρθει σε επαφή με την Θέρμη που είναι, όπως σας έλεγα, η Ισπανική Οργάνωση Εκπροσώπησης όλων των ανθρώπων με αναπηρίες στην Ισπανία. Δεν ξέρω αν συμφωνείτε, συνάδελφοι, γιατί δεν ήθελα ε, να παρουσιάσω μια δική μου πρωτοβουλία ως πρωτοβουλία της Επιτροπής. Τέλο πάντων αυτές είναι οι προτάσεις. Και εδώ ολοκληρώνουμε με την μίσια διάταξη. Η επόμενη συνεδρίαση είναι 11 Νοεμβρίου, 3 η ώρα το απόγευμα. Σας ευχαριστώ πολύ.